Right. Um, we, we had... Right, we better start, um, although there are not very many of us. Θα ξεκινήσουμε παρότι δεν είμαστε και αρκετοί. Θα ξεκινήσουμε με το σημείο το σημείο 8 εισηγητής για τους λογαριασμούς για το περιβάλλον είναι εισηγητής ο Χάνς Πέτερ Μάρτιν. Έχετε το λόγο, Χάνς Πέτερ. Καλή σας μέρα. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μου ερώτησε τι θα γίνει με τις προτάσεις μου. Δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί τη στιγμή που με ρώτησε ε, ήμουν ο μόνος στην αίθουσα εκτός από εσά πρόεδρε και είπα ότι οι προτάσεις μου θα τύχουν μια σερβιτά της πλειοψηφίας. Επιτρέψτε μου λοιπόν να κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις επίπεδο αρχής. Ε, καλύτερα μάλιστα που δεν είναι κανείς εδώ και δεν θα με ακούσουν πολλοί και δεν θα κάνω το λάθος που κάνουν πολλοί καθολικοί ιερείς, δηλαδή θεωρεί κανείς υπόλογους ε, κυρίως εκείνους που δεν επισκέπτονται την εκκλησία. Με πάση περιπτώσει, ερχόμενο εδώ σήμερα το πρωί σκεπτόμουν ότι θα είναι μία από αυτές τις ε, κλασικές στιγμές όπου συνάδελφοι θα ρωτήσετε μετά γιατί αυξάνεται η αγανάκτηση κατά της ε, πολιτικής, γιατί διευρύνεται η απόσταση ανάμεσα στους πολίτες και τους ερετούς ή και μη ερετούς εκπροσώπους που εμφανίζονται μέσω καταλόγων. Σήμερα λοιπόν το πρωί ε, θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω τη δική μου άποψη από αυτού. Σε εμά λοιπόν, όσον αφορά την πολιτική, υπάρχει κάτος, κάτι το οποίο είναι εξυπαρχής λάθος. Και είναι το εξής, ότι τελικά δεν κάνουμε εκείνο το οποίο περιμένουν από μας οι εκλογείς. Ε, και σε αυτό τι εννοώ, ε, για την προοπτική, για τις ε, ηγετικές ικανότητες, για την καθοδήγηση που ακριβώς θα μπορούσε να στραφεί μια εύρυθμα λειτουργούσα Ευρωπαϊκή Ένωση. Να υπάρχει ένα καλύτερο μοντέλο σε σχέση με τα υπόλοιπα να δούμε πού ακριβώς είναι τα πλεονεκτήματά μας, πού βρισκόμαστε λόγω της ιστορίας μας, πώς έχουμε προχωρήσει, βεβαίως και έχουμε και μειονεκτήματα και στην πραγματικότητα ποια είναι τα ουσιαστικά στοιχεία εκείνης της ε, άποψης ε, την οποία τρέφει η νέα γενιά ε, απέναντι στους πολιτικούς, κάτι το οποίο ενδεχομένως θα μπορούσε να τους ενδιαφέρει. Εγώ λοιπόν είμαι πεπισμένος ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα όπου αφενός οι κοινοβουλευτικοί, εμείς οι βουλευτές καλούμεθα και είμαστε σε μεγάλο βαθμό υπόλογοι, από την άλλη Όμω και μιλάω, επιτρέψτε μια παρένθεση, μιλάω πολύ αργά για να το καταλάβει και ο Πιέρ Λαμπέρ, κάτι με ενδιαφέρει πάρα πολύ, κλείνει η παρένθεση. Ε, να υπάρχει λοιπόν η ευκαιρία να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από την Ευρώπη. Out of Africa ως ε, κλισέ ας πούμε. Εσείς ε, κυρία Πρόεδρε, πολύ σωστά Είπατε σε μία από τις ε, τελευταίες ε, συνεδριάσεις ότι κανείς δεν πιστεύει πόσο σημαντικά είναι τα στατιστικά δεδομένα. Στη δική μας την Επιτροπή γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα στατιστικά στοιχεία σε κάποιο βαθμό ήταν ε, ενοχλητικά. Εγώ βεβαίως ως ανεξάρτητος ε, ε, μπορούσα να συμμετέχω στην εντράση των συντονιστών και είχα την ευκαιρία να δω ε, τι γίνεται με όλο αυτό το, τον καταιγισμό των στατιστικών δεδομένων. Όμως με τη Eurostat διαπιστώσαμε ότι οι βάσεις της δουλειάς μας κατά κανόνα είναι τα δεδομένα τα στοιχεία. Και αν δεν μπορούμε να βασιστούμε στα στοιχεία, διότι θεωρούμε ότι είναι ε, ελλειπή, τότε παρουσιάζεται ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο μπορεί να στοιχείσει μερικές φορές και 300 δις ή και περισσότερο και προφανώς εδώ αναφέρομαι στην Ελλάδα. Περνάω τώρα λοιπόν στην ε, θέση μου. Θεωρώ ότι αυτή η δική μου παρέμβαση σήμερα είναι μια κλασική περίπτωση για το Κοινοβούλιο, για τους πεπισμένους Ευρωπαίους που επιθυμούν να έχουν μια προοπτική. Ας δούμε λοιπόν τι καταλάβαμε. Καταλάβαμε ότι ο μέχρι τώρα ορισμός της ευμάριας του well-being, βασίζεται ή βασιζόταν μόνο στα στοιχεία ανάπτυξης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και αυτό ήταν λάθος, διότι μπορούμε στον ε, στενό μας προσωπικό κύκλο να διαπιστώσουμε ότι αν δεν περάσουμε στην ποιοτική ανάπτυξη δεν θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι ακριβώς σημαίνει ανάπτυξη. Παράδειγμα, εγώ μεγάλωσα στην περιοχή Μπούντζε και εκεί είχαμε σχεδόν πάντα χιόνι ε, με πολύ μικρές ε, εξαιρέσεις. Υπάρχουν και εικόνες που το μαρτυρούν αυτό, όμως τώρα πια δεν έχουμε χιόνι ίσως ε, διότι υπάρχει η υπερθέρμανση του πλανήτη αλλά και διότι έχουν αλλάξει και οι κλιματικές συνθήκες. Που τι σημαίνει αυτό σήμερα στη δική μου την περιοχή για να απολαύσω χιόνι θα πρέπει να διανύσω μια απόσταση τουλάχιστον 100 χιλιόμετρων να έχω όλες τις δαπάνες μεταφοράς για να μπορώ να κάνω σκι. Αυτές όμως οι εξελίξεις κατ' ουσίαν παρουσιάζονται ως ε, ανάπτυξη διότι το αυτοκίνητό μου είναι πιο μεγάλο, διότι πληρώνω βενζίνη που έχει αυξηθεί, άρα δηλαδή υποτίθεται αυξάνεται η οικονομία στην περιοχή μου, στον Μπούντζε, μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη, αλλά με ποιο τίμημα. Η Κομισιόν μετά από πολλές προσπάθειες ε, ε, ε, κυρίως και μετά από παρεμβάσεις ΜΚΟ, ενεργών πολιτικών, ακαδημαϊκών και άλλων. Δεν ξέρω ποιος επιλήθηκε του θέματος αυτού στα τελευταία 5-6 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εν πάση περιπτώσει τώρα θα είχαμε την ευκαιρία να πούμε ναι πράγματι καταλάβαμε. Ναι πράγματι επιθυμούμε να κάνουμε άλλο ένα βήμα πιο πέρα. Δεν θέλουμε να βασιστούμε μόνο στην οικονομική κρίση και στις εμπειρίες που έχουμε κάνει. Να βασιστούμε σε αυτά που λένε οι νέοι που λένε ότι εμείς την ευμάρεια την ορίζουμε διαφορετικά. Εμείς συμπεριλαμβάνουμε διάφορα οράματα, γεγονότα παραδείγματος χάρη, να δούμε τι ακριβώς ε, γίνεται με τους ε, Κινέζους ε, τι γίνεται με τις πυκνοκατοικημένες περιοχές στη Γερμανία. Κατά την άποψή μου όλα αυτά τα στοιχεία αναγκαστικά συμπεριλαμβάνονται σε μια νέα μορφή της ε, ποιότητας ζωής και της ε, πρόοδου στην Ευρώπη. Η Κομισιόν ε, κάνει μια προσέγγιση προς αυτή την, προς αυτή την κατεύθυνση. Βλέπετε λοιπόν, εγώ είμαι πεπισμένος ότι στους διάφορους τομείς μπορούμε να επεξεργαστούμε διάφορα μοντέλα τα οποία θα αντιμετωπίζουν τις κλιματικές αλλαγές, την ε, παροχή υπηρεσιών, εδώ αναφέρομαι στην ε, τροπολογία παριθμών 9, στους, ε, πλούτο, στις πλούτοπαραγωγικές πηγές, σε πάρα πολλά. Να είμαστε λοιπόν θαραλέοι, να πούμε ναι, θέλουμε αυτή την προσέγγιση που να είναι πολύ πιο προχωρημένη από αυτή των κρατών μελών. Έτσι μόνο θα φτάσουμε κάπου και αυτό στοιχίζει χρήματα. Εγώ λοιπόν στηρίζω αυτή την προσέγγιση, διότι πιστεύω ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς υπάρχουν αρκετοί υπάλληλοι οι οποίοι μπορούν κάλλιστα να μεταταγούν στη Eurostat. Και διότι είμαι πεπισμένος ότι κάτι το τόσο βαρετό όπως είναι τα στατιστικά δεδομένα, αυτό το βαρετό είναι καθοριστική σημασία για τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Thank you very much. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λούντβικσον Σκιώδης. Θα ήθελα να σας πω ότι θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ε, ότι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μία νομική βάση για θέματα προπολογισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό έπρεπε να το έχουμε κάνει πολύ νωρίτερα. Ελπίζω λοιπόν ότι τώρα πλέον θα επιταχύνουμε κατά τη τις ε, Το θέμα δεν είναι όλα αυτά να τα τακτοποιήσουμε οριστικά. Το θέμα είναι ότι τώρα πρέπει να κάνουμε το πρώτο βήμα. Η στρατηγική της Ευρώπης του 2020 αναφέρεται στην οικονομική ανάπτυξη, ε, σε μια συνειδητή περιβαλλοντική πολιτική και δεν νομίζω ότι αρκεί απλά να τροποποιήσουμε τη δυνατότητα πρόσβασης στα ταστιστικά δεδομένα. Χρειαζόμαστε μια ευρύτερη βάση που θα αναφέρεται και στα περιβαλλοντικά δεδομένα. Τα βελτιωμένα περιβαλλοντικά στοιχεία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας το θέμα του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και αυτά τα στοιχεία να τα συμπεριλάβουμε στις οικονομικές μας αναλύσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να επιτύχουμε αυτή την καθοριστική αλλαγή προσέγγισης της οικονομίας, να επιδιώξουμε την πράσινη ανάπτυξη. Αυτά τα στατιστικά δεδομένα είναι τεχνικής φύσεως, αλλά είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε την ε, προοπτική μας, την οικονομική προοπτική μας. Και από μια τέτοια ανάλυση που θα περιλαμβάνει τη διάσταση του περιβάλλοντος θα προκύψουν πάρα πολλά ωφέλη. Θα έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα του τι ακριβώς λειτουργεί, οποτεδήποτε λαμβάνονται πολιτικά μέτρα και τι δεν μπορεί να λειτουργήσει. Οι τροπολογίες τις οποίες κατέθεσε ο κύριος Μάρτιν, οι τροπολογίες αυτές ε, είναι ε, ιδιαίτερα θετικές. Ο κύριος Μάρτιν υπογραμμίζει ότι πράγματι είναι δυνατόν να συμπεριληφθεί η διάσταση του περιβάλλοντος. Ένα πράγμα βέβαια ακόμα πρέπει να συζητήσουμε το ότι το σύστημα για ε, στατιστικά δεδομένα διάρκειας, αυτό πράγματι πρέπει να δρομολογηθεί. Είναι ένας μακρύς δρόμος και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και κάτι άλλο, το πώς ακριβώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ανάγκη περισσότερων πλούτοπαραγωγικών πηγών και πόρων, διότι ε, υποβάλουμε μεγαλύτερες απαιτήσει απέναντι στα κράτη-μέλη, αλλά πρώτα απ' όλα θα πρέπει να τους πούμε επενδύστε στα καλύτερα στατιστικά δεδομένα. Αυτό είναι ο κανόνας. Και πρέπει να δούμε πώς ακριβώς ε, οι αναφορές για το περιβάλλον μπορούν να συμπεριληφθούν πρακτικά στη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι αυτό είναι το πλαίσιο, το απαραίτητο για την εφαρμογή της ε, στρατηγικής 2020. Ε, Κατά τα άλλα, θεωρώ ότι χρειαζόμαστε την αγαστή συνεργασία για να μπορέσουμε να εκπονήσουμε και μια ικανοποιητική έκθεση. Ευχαριστώ. Ε, Φιλίπ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω χωρίς να ευχαριστήσω το Χάνς Πέτα. Αλλά ε, θα ήθελα να συζητήσω για το ποιοι είμαστε εδώ και πόσοι είμαστε εδώ. Τώρα είμαστε σοβαροί γύρω από αυτή την υπόθεση. Αν βλέπουμε εδώ το πώς είναι παρόντες και αν οι παρουσίες ε, αντιπροσωπεύουν και ε, θα έλεγα αντανακλούν το βάρος που δίνουμε στο συγκεκριμένο θέμα, ανησυχώ. Ανησυχώ ιδιαίτερα γιατί δεν νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα προχωρήσουν τα πράγματα σωστά. Βέβαια θα μπορεί να πει κανείς ότι αποδίδει την απουσία αυτή στο ότι τα στατιστικά στοιχεία κάνουν τον κόσμο να βαριούνται. Είναι αλήθεια αυτό, αλλά είναι αλήθεια μόνο για αυτούς οι οποίοι θέλουν να ασκούν την πολιτική τους δραστηριότητα εκτός δεδομένων και αριθμών. Εγώ έχω μάθει το αντίθετο. Θεωρώ ότι πρέπει να βασιστούμε στα δεδομένα και τα συγκεκριμένα στοιχεία και μετά να προσπαθήσουμε να βρούμε διαφορετικές, ε, διαφορετικά θεμέλια στην δραστηριότητά μας στην πολιτική. Νομίζω ότι στην ουσία για να καταλάβει κανείς που βρίσκεται πρέπει να είναι σε θέση να προσμετρήσει ε, τις επιπτώσεις ε, της παρέμβασής του και ε, αν δεν το κάνει αυτό δεν θα είναι σε θέση να γνωρίζει αν αυτό το οποίο κάνει είναι θετικό ή όχι. Συνεπώς αυτές οι συζητήσεις που γίνονται για το αν θα πρέπει να ξεφύγουμε από τον περιορισμό του ΑΕΠ σαν παράδειγμα Πολλοί πιστεύουν ότι δεν έχουμε τα δεδομένα τα οποία απαιτούνται για να πετύχουμε κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει βρίσκω την έκθεση του Hans Peter πολύ ενδιαφέρουσα. Τον ευχαριστώ και για αυτά τα οποία έγραψε και για αυτά τα οποία είπε. Συμφωνώ σχεδόν 100% μαζί του. Και θα υποστηρίξουμε την πρότασή σου. Ένα σημείο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ λίγο όχι επί της ουσίας θα πείτε, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει εδώ ένα θέμα, το θέμα του κόστους. Πιστεύουν πολλοί ότι δωρεάν γεύμα δεν δίδει κανείς. Αν κάποιος θέλει πράγματι ουσιαστικά δεδομένα, στατιστικά στοιχεία έγκυρα, πρέπει να τα πληρώσει. Από μόνα τους δεν θα υπάρξουν. Υπάρχει λοιπόν εδώ ε, ένα κομμάτι των επενδύσεων που πηγαίνουν προς τη Eurostat να πάνε προς άλλες κατευθύνσεις διευρύνοντας τις στατιστικές βάσεις έρευνας. Θα πρέπει φυσικά το κόστος να είναι ελεγχόμενο αλλά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το επιχείρημα του κόστους για να μην προχωρήσουμε στη συλλογή των στοιχείων αυτών. Είναι πολύ πιθανό ότι θα πρέπει κάποια άλλα στοιχεία που είναι άχρηστα να σταματήσουμε να τα συλλέγουμε. Ένα τελευταίο σημείο σχετικά με έναν πίνακα στοιχείων ο οποίος θα πρέπει να είναι συνεκτικός, αποτελεσματικός και φυσικά να υπερβαίνει απλά του ΑΕΠ, των στοιχείων γύρω από το ΑΕΠ από την 1η Ιανουαρίου όταν θα γίνει ο πρώτος μακροοικονομικός έλεγχος στα πλαίσια του λεγόμενου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, διαρωτώ με αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συμπεριλάβει στον πίνακά της και κάποιες μετρήσεις κοινωνικές και περιβαλλοντικές. Προφανώς τα στοιχεία αυτά δεν θα είναι τόσο αξιόπιστα και σκληρά στοιχεία σε εισαγωγικά όπως τα στοιχεία που προέρχονται από λογιστικές διαδικασίες, οικονομικές λογιστικές διαδικασίες αλλά είναι ένα πρώτο βήμα το οποίο πρέπει να γίνει. Πρέπει να καταστήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ικανή έτσι ώστε από την 1η Ιανουαρίου του 2012 να είναι σε θέση να λάβει όλα αυτά τα στοιχεία εξίσου υπόψη. Χανς Πέτερ σε ευχαριστούμε και θα πρέπει όλοι εδώ να προσπαθήσουμε να συνειδητοποιήσουμε στα πλαίσια των πολιτικών μας ομάδων ότι το θέμα αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο βάρος. Βίκη Φόρντ. Ζητώ συγγνώμη που ήρθε καθυστερημένη, λέει προς τον Χάνς Πέτα. Υπάρχουν κάποιες πολιτικές ανησυχίες σχετικά με τον περιβαλλοντικό φόρο και την πλήρη εφαρμογή της αρχής ο αυτός που μολύνει είναι αυτός που θα πληρώνει επίσης. Υπάρχουν πάντως ε, νομίζω ιδέες ξεκάθαρες σχετικά με την χρησιμότητα των περιβαλλοντικών στοιχείων τα οποία θα μας επιτρέψουν να κάνουμε και ποσοτικά και συγκριτικά περαιτέρω αναλύσεις. Βέβαια δεν υπάρχει καθολικά αποδεκτό πρότυπο για την ποσοστικοποίηση τέτοιου είδους ε, περιβαλλοντικών μέτρων και ακόμα και σε επίπεδο ορολογίας υπάρχουν σημαντικές διαφορές θα θέλαμε εμείς να προσπαθήσουμε να συντονίσουμε τα δεδομένα και τους ορισμούς που χρησιμοποιούμε και με οργανισμούς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να αποφύγουμε κάποιες δυνατότητες διεκτησίας ή πλειοδοσίας καλύτερα αν θέλετε ανάμεσα σε διαφορετικά περιβαλλοντικά καθεστώτα. Εσείς προτείνετε να δώσουμε στη Eurostat ε, και συμφωνώ με αυτό ε, χρήματα πιστώσεις από υπάρχοντες, ε, από, από άλλες θέσεις του προϋπολογισμού. Λοιπόν, αυτά. Χάνς Πέτα, θες να δώσεις κάποια απάντηση. Σε ευχαριστώ που μου έδωσες ξανά το λόγο. Ευχαριστώ τα σχόλια για την ομιλία μου. Καλό θα ήταν αυτά που άκουσαν να αντικατοπτρίζουν την κοινή στάση της Επιτροπής μας γύρω από την προσπάθεια αυτή. Από το παρελθόν μου ως δημοσιογράφο νομίζω ότι πρέπει να πω ότι θα σταθούμε, πρέπει να σταθούμε θαραλέοι, θα πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα μας προς τα εμπρός και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τα ευρωπαϊκά δεδομένα για την αηφορία. Αν προσπαθήσουμε να τα ορίσουμε σωστά, τότε θα δώσουμε και προς τα έξω την εικόνα, η οποία θα επιτρέψει στον κόσμο να καταλάβει αυτά τα οποία προτείνουμε. Το θέμα της χρηματοδότησης θα πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω. Κατανοώ αυτά που είπε ο Λάμπερτς και αυτά που είπε η Φόρντ αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι το θέμα της χρηματοδότησης χρήζει περαιτέρω επεξεργασίας. Και νομίζω ότι τίθενται ορισμένα ερωτηματικά. Τόσοι και τόσοι υπάλληλοι, τόσες πιστώσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεύρυνση, σαν παράδειγμα. Πού είναι όλοι αυτοί, τι κάνουν σήμερα. Νομίζω ότι υπάρχει η δυνατότητα ένας αριθμός από τις θέσεις αυτές να μετακινηθεί προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση, συνοδευόμενη μετακίνηση αυτή από τα απαιτούμενα κονδύλια. Θα νομίζω ότι υπάρχουν κάποια τμήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ολοκλήρωσαν ε, την αποστολή τους και δεν θα πρέπει να συνεχίσουν να διαιωνίζονται. Ευχαριστώ. Το χρονοδιάγραμμα, η προθεσμία μάλλον για την κατάθεση τροπολογιών είναι η 1η Οκτωβρίου. Εξέταση τροπολογιών 18 Οκτωβρίου, ψηφοφορία 26 Οκτωβρίου, έτσι ώστε η επί της ουσίας Επιτροπή να τα εξετάσει στις 9 Δεκεμβρίου, Νοεμβρίου και να φτάσουμε ε, για ψηφοφορία στην Ολομέλεια στη 2η του Νοεμβρίου. Περνάω τώρα στο σημείο 9. Μέτρα για την προώθηση ε, της χρηστής διακυβέρνησης οικονομικής σε χώρες ε, τρίτες συνεργαζόμενες αναπτυσσόμενες χώρες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Ζητά συγγνώμη συγκήτρια που δεν μπορεί να είναι εδώ γιατί υπάρχουν ψηφοφορίες στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Θα μιλήσω λοιπόν εγώ εξ ονοματός της. Σε αυτό το σχέδιο της γνωμοδότησης <clears throat> χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Κομισιόν και αναγνωρίζει την ανάγκη να υπάρχει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο θα αφορά ε, στην οικονομική ανάπτυξη και στις εξελίξεις ε, στον ιδιωτικό τομέα. Επισημαίνει ότι προοδευτικά οι φτωχές ε, χώρες ε, πρέπει να αντικαταστήσουν την ε, εξωτερική βοήθεια με αποτελεσματικό φορολογικό ή δημοσιονομικό σύστημα. Γιατί υπάρχουν προσκόμματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Σε αυτήν λοιπόν τη γνωμοδότηση καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει πλέον αυστηρά κριτήρια για την αναγνώριση φορολογικών παραδείσων και να εργαστεί προς μια δεσμευτική, διεθνή, πολυμερή και αυτόματη συμφωνία ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών. Και τέλος, θεωρεί ότι οι αρχές της χρηστής διαχείρισης στον τομέα της φορολογίας ε, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε όλες τις συμφωνίες που συνάπτουν ε, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ίδια η Ένωση. Νομίζω ότι αυτά είναι τα τρία-τέσσερα βασικά στοιχεία στη γνωμοδότησή της. Ε, με μεγάλη μου χαρά ε, προσβλέπω στις ε, απαντήσεις σας και θα διαβιβάσω τις απόψεις σας στην ΣΥΡΠΑ. Η Βίκη ζήτησε το λόγο. Ζητώ συγγνώμη που και εγώ αντικαθιστώ τη συναδελφό μου που δεν μπορεί να είναι εδώ και μου ζήτησε να αναφέρω τα εξής. Είναι σημαντικό λοιπόν να εντοπίσουμε τα κριτήρια για να εντοπίσουμε του φορολογικού παραδείσου. Επίση όμω είναι σημαντικό να πούμε ότι οι αναπτυσσόμενε χώρε ε, πρέπει να προσπαθήσουν να εφαρμόσουν ένα ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα, ε, να κάνουν επενδύσει για του ε, αυτόχθονε. Είναι επίση σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η χαμηλή φορολόγηση δίνει τη δυνατότητα στο να υπάρχουν περισσότερε αγωγέ και στη τελική ανάλυση ε, μέσα από κάποιε αντισταθμίσει να υπάρχει ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα. Οι ειδικοί για τι αναπτυσσόμενε χώρε εκφράζουν ε, ανησυχίε για το ότι πολλέ από αυτέ ε, εξαρτώνται μόνο από την βοήθεια που λαμβάνουν, την αναπτυξιακή βοήθεια και δεν ασχολούνται με τα υπόλοιπα τα φορολογικά. Ο Σβέν. Πολύ σύντομα, ευχαριστώ και αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης πολύ καλά έχει συνταχθεί και πολλά από τα σημαντικότερα σημεία τα οποία συζητήθηκαν πολλές φορές συμπεριλαμβάνονται στις προτάσεις. Πιστεύω ότι τουλάχιστον στη γερμανική μετάφραση η αιτιολογική σκέψη 7 θα μπορούσε να γίνει καλύτερη διότι όπως είπαμε, δεν χρειάζεται να δημοσιεύουν σε ενιαία βάση οι εταιρείε τους οικονομικούς λογαριασμούς, αλλά κάθε μία θα πρέπει να το κάνει χωριστά. Και βεβαίως η φορολογία θα πρέπει να αντιστοιχεί με αυτό που ισχύει σε κάθε χώρα. Δεν θα πρέπει όμως να ξεχνούμε ότι αν μπούμε σε τέτοιου είδους λεπτομέρειες για αυτή τη συζήτηση, σε κάποιες περιοχές του κόσμου ήδη υπάρχει... Ε, γίνεται μεγάλη μάχη για τον φορολογικό ανταγωνισμό. Όπως είπε λοιπόν και η Βίκη, θα πρέπει να δούμε μέσω διακρατικής συνεργασίας ποιες είναι αυτές οι χώρες. Και όταν στις αναπτυσσόμενες χώρες υπάρχει αναπτυσσιακός φόρος 0%, τι γίνεται. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της πραγματικότητας και του ονομαστικού φόρου. Όταν είμαστε στην ε, πραγματικότητα ε, στο μηδέν, για πώς μπορεί κανείς να είναι ανταγωνιστικός. Θα πρέπει να το δούμε διαφορετικά. Το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι αναπτυγμένες χώρες δεν μπορούν να προσφέρουν έναν ίδιο με τρίου ύψους ε, φόρο αν θέλετε, διότι υπάρχει μεγάλη ανταγωνιστικότητα. Θα πρέπει λοιπόν ό,τι κάνουμε να το δούμε με ισοσκελισμένο τρόπο και να μην έχουμε μόνο τέτοιου είδους ανταγωνιστικά επίπεδα φορολογικά τα οποία ισχύουν μόνο για ολίγους. Βλέπω να θέλει κανείς άλλος να λάβει το λόγο. Θέλει κανείς να... Θέλετε να επανέλθετε. Ε, σας ευχαριστώ για τα σχόλια και θα τα μεταφέρω στην ΣΥΡΠΟ. κύριος Λάμπερτ. Θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Στην έκθεση αναφέρεται η αναφορά για κάθε χώρα χωριστά. Πιστεύω ότι αυτή η υποχρέωση θα πρέπει να ισχύει για όλες τις εταιρείε οι οποίες ε, ε, δραστηριοποιούνται διακρατικά. Δεν αναφέρεται το σφαιρικό ευθυτή. Πάντα όταν το αναφέρουμε λέμε θα πρέπει να είναι συνολικό ή όχι. Δεν βλέπω γιατί θα πρέπει να μην το συζητήσουμε αυτό και αυτό ίσως θα πρέπει να αναφερθεί. Σας ευχαριστώ. Η συντάκτρια της ε, γνωμοδότησης θα λάβει υπόψη τα σχολεία σας. Περνούμε στο επόμενο θέμα. 10. Χορήγηση εγγύηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από δάνεια και εγγύηση στα σχέδια εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιμένουμε τον ε, συντάκτη τη γνωμοδότηση. Κυρία Σάι, θα ήθελα να μου εξηγήσετε τις προθεσμίες για την προηγούμενη έκθεση. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών, 4 Οκτωβρίου. 26 Οκτωβρίου θα τις εξετάσουμε, θα ψηφίσουμε στην οίκον στις 8 Νοεμβρίου, ώστε η επί της ουσίας, πέφτηνη η Επιτροπή, η ΕΝΒΗ, όχι, η ΤΕΒΗ Ανάπτυξη, ε, να τις έχει έτοιμες, διότι θα τα ψηφίσει στις 9 ε, Δεκεμβρίου. Περιμένουμε λίγα λεπτά να έρθει ο συντάκτης της επόμενης γνωματότητας. Το πρόβλημα είναι ότι κάνει την παρουσίαση μιας άλλης ε, ε έκθεσης σε μια άλλη επιτροπή πολλές φορές συμπίπτουν. Right. Um, σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Θα συνεχίσουμε τώρα. Όπως σας εξήγησα προηγουμένως, ο εισηγητής έχει μεγάλη ζήτηση, ήταν σε πολλές επιτροπές, αλλά θα μας μιλήσει τώρα για τις εγγυήσει προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων όταν υπάρχουν ζημίες από ε, δάνεια εκ εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει το λόγο ο κύριος Κούτας. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη για την καθυστερημένη έλευση. Αλλά έχω και άλλη μια έκθεση σε άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή. Τα στοιχεία γύρω από τη νέα πρόταση απόφασης νομίζω ότι είναι γενικά θετικά ενισχύουν την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να υποστηρίξει τις νέες αναπτυξιακές δραστηριότητες, αυξάνουν τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στον τομέα των υποδομών για το περιβάλλον και τις συγκοινωνίες και τις μεταφορές, όπως επίσης και τη συμμετοχή της σε έργα τα οποία έχουν σαν στόχο την μετρίαση θα λέγαμε των επιπτώσεων της υπερθέρμανσης της ατμόσφαιρας του κλίματος. Υπογραμμίζεται επίσης ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα πλαίσια της νέας οικονομικής δραστηριότητας, η καταπολέμηση της, απασχ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων διασφαλίζει ότι οι στόχοι οι οποίοι περιλαμβάνονται στην απόφαση αυτή θα γίνονται σεβαστοί σε όλα τα προγράμματα στα οποία θα εμπλακεί. Υπάρχει ανάγκη για παγκόσμια, για σφαιρική, δημοσιονομική, συγγνώμη, χρηματοπιστωτική συνεργασία και φυσικά πρέπει να υπάρξει ειδική αντιμετώπιση των περιοχών οι οποίες χαρακτηρίζονται ή των χωρών οι οποίες χαρακτηρίζονται σαν φορολογική παράδειση. Για να συνεχιστεί και η συμφωνία η οποία έχει υπάρξει μέχρι τώρα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τα άλλα θεσμικά όργανα θα πρέπει να υπογραφεί και η νέα αυτή σύμβαση. Σας ευχαριστώ και περιμένω τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ πολύ λέει η Πρόεδρος. Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει το λόγο. Ο Σβέν έχει ζητήσει το λόγο. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Προϋπολογισμών το καλό σχέδιο γνωμοδότησης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Κούτας για τις καλές προτάσεις που υποβάλλει για να γίνουν συμπληρωματικές αλλαγέ. Μόνο λίγες παρατηρήσεις. Βεβαίω δεν είμαστε αντίθετοι με οποιαδήποτε από τι ιδέε που εκφράζονται και τι προτάσει. Θα θέλαμε όμω να γίνουν κάποιε συμπληρωματικέ αλλαγέ. Μία από τι οποίε είναι στο σημείο 7 και αν δεν κάνω λάθος στο σημείο 9 που δίδεται ο ορισμός των φορολογικών παραδείσων που βασίζεται στους καταλόγους του ΟΣΑ. Είναι όμως κενός αυτός ο ορισμός. Είναι τόσο αστείος αυτός ο ορισμός που κατά κάποιο τρόπο κάνει όλους τους φορολογικούς παραδείσους να εξαφανίζονται. Αυτό όμως δεν είναι αληθές θα πρέπει στα κριτήρια του καταλόγου να προσθέσουμε ότι όταν γίνει αποτελεσματική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στην Ευρώπη, θα δούμε ποιες είναι οι χώρες που δεν συνεργάζονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρούνται ως φορολογική παράδοση, διότι είναι αστείο αυτό με τον κατάλογο των φορολογικών παραδείσων στον οποίο δεν υπάρχει καμία χώρα Δεύτερον, πιστεύουμε ότι καλό είναι η ΕΤΕΠ να κάνει πιο αποτελεσματική και καλή χρηματοδότηση, αλλά θα πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι πολλές φορές χρηματοδοτούν και μη αηφόρα σχέδια. Θα βάλουμε θα υποβάλουμε ούτω ή άλλω γραπτό προτάσει μα για περαιτέρω τροπολόγηση σε σχέση αυτά που ανέφερα και θα τα συζητήσουμε ώστε να μπορέσουμε στο τέλος να έχουμε μία πρόταση με την οποία θα συμφωνήσει η μεγάλη πλειοψηφία των μελών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πιστεύω ότι είναι ενδιαφέρουσα η ιδέα να κάνουμε κάτι για τον ορισμό των φορολογικών παραδείσων. Αλλά διερωτώ εάν μπορούμε να ακολουθήσουμε την πρόταση του Σφέντς. Όντως, ε, πρόκειται για κάτι το ε, ουτοπικό, αλλά ακόμη δεν είναι κάτι το οποίο έχει ακόμη γίνει αποδεκτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δύσκολο να ζητούμε να το κάνουν κάποιοι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν εμείς δεν μπορούμε να κανονίσουμε, να νοικοκυρέψουμε τα του οίκου μας. Δεν έχω πρόταση, λέει πρόεδρος, απαντώντας στον Σβέν. Ίσως όμως θα μπορούσα εγώ να δω ένα νέο ορισμό το πνεύμα της ε, παρατήρησής σας με βρίσκει σύμφωνη, αλλά ίσως θα πρέπει να πούμε ότι ίσως ο απότερος αντικειμενικός στόχος είναι αυτό, δηλαδή να έχουμε ε, κάποιον σε, αυτή την, ε, σε αυτό τον κατάλογο των φορολογικών ε, παραδείσων. Προς το παρόν δεν υπάρχει κανείς, αλλά ίσως αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλεται και στο επίπεδο ακόμη της τεχνολογίας και αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να κάνουμε σιγά σιγά κάποια βήματα για να βελτιωθεί η κατάσταση. Ο κύριος Κούτας, ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν ξέρω αν υπάρχει εκπρόσωπος της τράπεζας εδώ. Είχαμε... Έχουν γίνει ήδη κάποιες συζήτησεις. Αν είναι εδώ θα μπορούσαν να μας πούνε τις ιδέες τους. Ευχαριστώ τον συνάδελφο και είμαι ανοιχτό σε οποιαδήποτε υπόδειξη. Και θα ήθελα και εγώ να βρούμε μια λύση για τον ορισμό αυτών των φορολογικών παραδείσων. Όπως είπατε, και εγώ είμαι έτοιμος να συζητήσω με τον οποιοδήποτε για να ευρεθεί λύση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα έχουμε βεβαίως την ε, δυνατότητα σε 10 λεπτά να κάνουμε ερωτήσεις ο κύριος Στολογιάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχει σχέση με την έκθεση αυτή η ερώτησή μου, αλλά με τους φορολογικούς παραδείσους. Θέλω να σας πω ότι για τους πολίτες που ζουν στις χώρες μας, πιστεύω ότι θα πρέπει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να το σκεφτούν πάρα πολύ σοβαρά το θέμα αυτό. Υπάρχει μία πρόταση η οποία πολλές φορές εμφανίζεται μπροστά μας, που απορρίπτεται πάντα. Αλλά πρόκειται για μία πρόταση που υποστηρίζουν οι πολίτες μας. Και είναι η εξής. Υπάρχουν χώρες στις οποίες, οι οποίες είναι φορολογική παράδοση και δεν συμφωνούν να έχουν καμία συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για λόγους διαφάνειας. Και διαρωτώ με αν δεν θα πρέπει να σταματήσουν τις δραστηριότητες τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι εταιρείε που έχουν εγγραφεί και έχουν την έδρα τους σε φορολογικούς αδρήμες και δεν ε, υπογράφουν συμφωνίες διαφάνειες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα μέτρο που κατά κάποιο τρόπο θα ανταποκριθεί στα αιτήματα των ε, πολιτών μας. Διότι όντως υπάρχουν πολλές εταιρείες οι οποίες είναι, έχουν την έδρα τους σε τέτοιου είδους φορολογικούς παραδείσους, κάνουν ε, συναλλαγές, ε, αλλάζουν την ιδιοκτησία της εταιρείας, δίζουν πάρα πολλά χρήματα και οι χώρες στις οποίες δραστηριοποιούνται δεν μπορούν να τις φορολογήσουν. Και αυτό νομίζω ότι δεν είναι έντιμο, δεν είναι δίκαιο. Ο Σβέν. Νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να πάμε. Όντως, μπορεί κανείς ε, να σκεφτεί ποιες είναι οι κυρώσεις που μπορούν να εφαρμοστούν, αλλά θα, υπάρχει να θα πρέπει να υπάρχει κάποια κύρωση. Συμφωνώ πλήρως, τουλάχιστον στη Γερμανία, σύμφωνα με τον νόμο προβλέπονται κυρώσεις για οποιαδήποτε μεταφορά χρημάτων γίνεται προς φορολογικούς παραδείσους. Το πρόβλημα είναι ότι ο κατάλογος των φορολογικών παραδείσων βασίζει τον κατάλογο του ΟΣΑΠ, όπως είπα δεν περιέχει κανένα φορολογικό παράδεισο, είναι άδειο. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να κάνουμε τον ορισμό του και μετά να προβλέψουμε ποιες είναι οι κυρώσεις. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε κάποιες χώρες να καταχρώνται τις ε, κεφαλικές ε, αγορές ε, και τις ανοιχτές αγορές εξαιτίας των φορολογικών παραδείσων. Διότι ο φορολογικός παράδεισος δεν είναι, μοιάζει με τον παράδεισο τον κανονικό. Ο παράδεισος είναι μια πολύ σημαντική λέξη δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα οποία γίνονται σε αυτούς τους φορολογικούς παραδείσους. Ακούστε, ο φορολογικός παράδεισος είναι παράδεισος για κάποιους. Περί αυτού πρόκειται, λέει η Πρόεδρος. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αυτή είναι μια γενικότερη συζήτηση. Μπορούμε να επιβάλλουμε στον κύριο Κούτα να τη συμπεριλάβει στην έκθεση του. Και στην έκθεση Ντομινιτσί, αν θυμάστε, Είχαμε προβλέψει κάτι, αλλά δεν υπερψηφίστηκε. Ίσως θα μπορούσαμε την επόμενη φορά ε, στις διάφορες σχετικές εκθέσεις να προχωρήσουμε πιο προοδευτικά. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα έχουμε πέντε λεπτά στη διάθεσή μας πριν να ακούσουμε τον ε, επόμενο μιλητή. Λοιπόν, το χρονοδιάγραμμα κατάθεση τροπολογιών έως την 1η Οκτωβρίου. Εξέτασή τους στις 18. Ψηφοφορίες στην Επιτροπή μας 26 Οκτωβρίου. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθήσουμε. Right. Um, σα ευχαριστώ συνάδελφοι. Περνάμε στο σημείο 11 της ημερήσιας διάταξης ανταλλαγή απόψεων με τον Φιλίπ Μεστάτ, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και πρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου. Θα ήθελα να μας παρουσιάσει ο κύριος Μεστάτ τα πεπραγμένα της τράπεζάς του τον τελευταίο χρόνο και για τον ρόλο που μπορεί να παίξει η τράπεζα αυτή συμπληρώνοντας τον κοινοτικό προϋπολογισμό σε μεγάλα επενδυτικά προγράμματα στο μέλλον. Ξέρετε ότι υπάρχει και μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για την ετήσια σας έκθεση. Η συγητής μας είναι ο κύριος Κούτας. και θα είναι ο πρώτος ο οποίος θα ξεκινήσει με ερωτήσεις αφού φυσικά κύριε Μεστάτ σας ακούσουμε. Thank you very much. La ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε να σας μιλήσω για τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεως. Σε αυτές τις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις θα αναφερθώ και δύο στις δραστηριότητες της ΕΤΕ εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω είπε και η πρόεδρο, θα... το οποίο πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να συνεισφέρουμε με τι δραστηριότητέ μα στι οικονομικέ τη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα κάνω δύο εισαγωγικέ παρατηρήσει. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να υπογραμμίσω την εξαιρετική συνεργασία που έχω με την Επιτροπή σα. Όπω ξέρετε, σύμφωνα με τι συνθήκε, η Ευρωπαϊκή Τραπέζα Επενδύσεων δεν είναι υπόλογη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκτιμώ όμως ότι αυτό εξυπακούεται και είναι κάτι το οποίο επιβάλλεται φυσικό το τρόπο, δεδομένου ότι είμαστε ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο στην υπηρεσία των ευρωπαϊκής πολιτικής γενικότερα. Είναι λοιπόν απόλυτα φυσιολογικό να είμαι θα υπόλογη και να κάνουμε αναφορά σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Θα ήθελα να σας πω ποια είναι ε, τι ακριβώς έγινε ε, ε, για την, εφαρμογή των φάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μετά στη θέση σας. Δεύτερη συλλογική παρατήρηση είναι ότι σήμερα στην ημερήσια διάταξή σας εξετάζεται και το θέμα της εξωτερικής, των εξωτερικών δραστηριοτήτων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης της ΕΤΕ και αν έχετε ερωτήσεις για αυτό το θέμα είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαρίστω θα απαντήσω. Ποιο είναι λοιπόν ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ο ρόλος μας στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης. Όταν ξέσπασε το τέλος του 2008 η οικονομική κρίση, οι μέτοχοι μας, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας ζήτησαν να αυξήσουμε όσο περισσότερο μπορούσαμε την υποστήριξή μας προς ε, διάφορα σχέδια, να αυξήσουμε τα δάνεια που χορηγούμε προς τρεις κατευθύνσεις, κυρίως προς τις ε, χώρες, τις περιοχές σύγκλησης, κλιματική αλλαγή και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γνωρίζετε τους αριθμούς για το 2009. Υπογράψαμε δάνεια της τάξεως των 79 δις ευρώ, δηλαδή είχαμε 37% αύξηση το 2009 σε σχέση με το 2008 και 66% σε σχέση με το 2007. Ήταν λοιπόν ουσιαστική η αύξηση του ε, όγκου των δραστηριοτήτων μας. Από αυτά 29 δις πήγαν σε project που ε, σε περιοχές σύγκλησης, 17 σε σχέδια που συνεισφέρουν άμεσα στην μείωση ε, των ε, εκπομπών διοξιδίου και 12 διατέθηκαν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω των πιστοτικών ιδρυμάτων με τα οποία συνεργαζόμαστε. Πάρα πολύ σύντομα λοιπόν, αυτό συνέβη το 2009. Το ερώτημα είναι πώς μπορούμε τώρα να επαναπροσδιορίσουμε τις δράσεις μας για το μέλλον. Λαμβάνουμε υπόψη κυρίως δύο στοιχεία. Αφενός το ότι ευτυχώς υπάρχει μια κάποια ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρώπη. Ακόμη είναι ευάλωτα τα πράγματα, αλλά βεβαίως βλέπουμε σιγά σιγά να επιβεβαιώνεται αυτή η ανάκαμψη μετά και από την αύξηση των εξαγωγών και τα πρώτα δείγματα αύξησης της εσωτερικής ε, ζήτησης άλλες χώρες μας, τι σημαίνει ότι εμείς έχουμε κάποιους πελάτες, αν θέλετε, που χρειάστηκε να υποστηρίξουμε το 2009, οι οποίοι έχουν λιγότερο ανάγκη από την ΕΤΕ το 2009. Πρόκειται για τις μεγάλες εταιρείε και επιχειρήσεις. Από το σύνολο των 79 δις του 2009, το 42% πήγαν προς επιχειρήσεις, δηλαδή ποσοστό υψηλότερο του συνήθους, αλλά είχαν προβλήματα χρηματοδότησης το 2009 αυτές οι εταιρείες διότι είχαν πολύ περισσότερους ε, ενδιασμούς οι τραπεζίτες στους οποίους απευθύνονταν συνήθω. Υπάρχει βελτίωση το 2010 και τόσο το καλύτερο, διότι ή ε, απευθύνονται απευθεία στην κεφαλαία χώρα πλέον ή προς τους συνήθεις χρηματοδότους τράπεζας. Ένα μέλος των πελατών μας, λοιπόν, αυτοί οι πελάτες, οι εταιρείε χρειάζονται λιγότερα, αλλά μπορούμε να μειώσουμε τον όγκο των ε, δανείων μας προς αυτές. Ένα δεύτερο στοιχείο πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι το γεγονός ότι δεν μπορούμε επί πολλά συνεχεία να έχουμε τόσο υψηλό επίπεδο δραστηριοτήτων, διότι καταναλώνουμε κεφάλαιο και θα φτάσουμε στο ανώτατο όριο, έτσι όπως το ορίζει το καταστατικό μας που είναι παράρτημα των συνθήκων. Εκεί προβλέπεται ότι το σύνολο των ε, τρεχόντων, τρε, συγγνώμη, τρεχουσών δραστηριοτήτων μας δεν μπορεί να ξεπεράσει το 250 του συνολικού μας κεφαλαίου. Και αν ζητήσουμε αύξηση του κεφαλαίου, θα μας πούνε οι μέτοχοι να το κάνετε από τη στιγμή που δεν θα κοστίσει αυτό ούτε ένα ευρώ στους κρατικούς μας προϋπολογισμούς. Πράγμα σημαίνει ότι θα πρέπει να αυτοχρηματοδοτήσουμε την αύξηση του κεφαλαίου και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε αρκετό χρόνο για να δημιουργήσουμε αποθεματικό βάσει των ετησίων κερδών μας για να μπορούμε να αυτοχρηματοδοτούμε την αύξηση του κεφαλαίου αν θέλουμε. Και αυτό βεβαίως δεν μπορεί να γίνεται για πολλά συνεχή έτη. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να προσανατολίσουμε τις δραστηριότητες μας προς τομείς στους οποίους η δράση μας, θα είναι πιο ενδιαφέρουσα. Γι' αυτό σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθούμε να δούμε σε ποιο μέτρο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί να συνεισφέρει στην ε, εφαρμογή της στρατηγικής 2020. Πιστεύω ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσει εφαρμογή αυτή τη στρατηγική. Είμαι πεπισμένο ότι πρόκειται για την ε, ορθή στρατηγική και είναι πρωταρχική σημασία για τους Ευρωπαίους να αυξήσουν το δυναμικό αύξηση. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα πρέπει να αυξηθεί η παραγωγικότητα, τι σημαίνει επίσης αυτό, ότι θα πρέπει να γίνουν μεγαλύτερες προσπάθειες σε θέματα κατάρτισης, έρευνας, ανάπτυξης και εκτιμώ ότι συνδυάζοντας τις δράσεις με αυτές Τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούμε να συνεισφέρουμε στη θέση εφαρμογή αυτή τη στρατηγική. Και ποια είναι τα θέματα που συζητούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τρόποι που θα μας επιτρέψουν με δάνεια της ΕΤΕ να δώσουμε με τα ίδια μέσα του προϋπολογισμού μια νέα όθηση και να κάνουμε κάτι το καλύτερο, κάτι περισσότερο βασιζόμενοι είπα σε αυτά τα δάνεια. Και σε θέματα κεφαλαίου να ελαφρύνουμε το άχθος για την ΕΤΕ. Αν λοιπόν δεν συνεργαστούμε με την Κομισιό, οι περιορισμοί που έχουμε μετά τη συμφωνία της Βασιλείας 3 σημαίνει ότι θα εξαντλήσουμε το κεφάλαιο που διαθέτουμε πιο σύντομα. Σε συνεργασία λοιπόν επαναλαμβάνω με την Κομισιό έχουμε μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Ένα παράδειγμα το Risk Finance Research Facility για τα θέματα της έρευνας. Με λίγα λόγια. Θέτουμε από κοινού μέσα από τον ε, κοινοτικό προπολογισμό, από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και οικονομικούς πόρους της ΕΤΕ. Ένα δις, το οποίο πήραμε από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και ένα δις από τα κέρδη της ΕΤΕ. Έτσι, κάνουμε ένα αποθεματικό που μας επιτρέπει να δανείζουμε περισσότερο για ε, δραστηριότητες κινδύνου ή για project τα οποία σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης είναι σημαντικά και μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο, διότι έχουμε αυτό, όπως σας είπα, το αποθεματικό. Αυτό το μαξιλαράκι που έχουμε δημιουργήσει, που μας επιτρέπει να ενεργούμε καλύτερα. Αυτά λοιπόν τα δύο δις που έχουμε βρει από κοινού, μας επιτρέπουν να δανείζουμε ποσά που συνολικά είναι πάνω από 10 δις. Εμείς βεβαίως ε, χρηματοδοτούμε εν μέρη τέτοιου είδους ε, δραστηριότητες και αυτό είναι ένας μοχλός αν θέλετε που μας βοηθάει. Και βεβαίως πρόκειται για μια δραστηριότητα που είναι ενδιαφέρουσα και για μας, γιατί αν κάναμε μόνοι μας αυτή την επικίνδυνη χρηματοδότηση θα δεσμεύαμε πολύ περισσότερο τα δικά μας κεφάλαια. Και εδώ, επειδή μοιραζόμαστε το ρίσκο, εφόσον λέγεται αυτό risk sharing με την Κομισιό, είμαστε σε καλύτερη ε, κατάσταση αν θέλετε. Επίσης, από κοινού με την Κομισιό επεξεργαζόμαστε τέτοιου είδους μέσα στα πλαίσια κάποιων κριτηρίων. Δηλαδή, τέτοιου είδους σχέδια θα πρέπει να είναι απλά, Γι' αυτό πάντα με την Κομισιόν διαπραγματευόμαστε ένα, ε, μια συμφωνία πλαίσιο για αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα. Δεύτερον, θα πρέπει να είναι revolving, δηλαδή εάν, ε, να έχουν κάποια απόδοση, εάν όλα πάνε καλά, ανακτούμε ένα χρήμα ένα μέρος των χρημάτων που δώσαμε και μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε κάποιο άλλο σχέδιο. Και τρίτον, αυτά τα μέσα θα πρέπει να είναι καταλυτικά, όπως τα ονομάζουμε. Δηλαδή, να είναι η ευκαιρία να μπορέσουμε να, να ε, προσελκύσουμε προς εμάς άλλα χρηματοδοτικά μέσα από το, δημοτικό, από το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Θα πρέπει να κάνουμε δηλαδή κάτι το ελκυστικό. Ο πρόεδρος Μπαγόζο στο μήνυμά του για την κατάσταση ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση σας μίλησε και για τα project bonds, για κάποιο άλλο μέσο. Η οικονομική κρίση, όπως ξέρετε, είχε αρνητικές επιπτώσεις στο project finance στις περισσότερες χώρες μέλη. Αυτή με χρηματοδότηση γεννηδότερα των κρατών μελών, τα οποία έχουν τους οικονομικούς περιορισμούς που γνωρίζετε. Απ' την άλλη, οι ανάγκες για έργα υποδομής είναι εξαιρετικά σημαντικές για τις επόμενες δεκαετίες. Πριν από την κρίση κατορθώναμε να, να κινητοποιήσουμε ιδιωτικά κεφάλαια διότι οι επενδυτές, οι μακροπρόθεσμοι, δηλαδή συνταξιοδοτικά ταμεία ή ασφαλιστικά ταμεία, αγόραζαν ομόλογα στα πλαίσια των έργων υποδομής που είχαμε προβλέψει. Αυτά τα ομόλογα είχαν καλή απόδοση διότι υπήρχε εγγύηση από τις monolines όπως λέγουμε. Με την κρίση οι monolines εξαφανίστηκαν, αυτό το μέρος της αγοράς εξαφανίστηκε και είπαμε την Κομισιόν πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι για να προσελκύσουμε και πάλι τα ιδιωτικά κεφάλαια για να χρηματοδοτούμε τέτοιου είδους ε, ε, σχέδια για έργα υποδομής. Αυτό λοιπόν, έτσι καταλήξαμε στα project bonds. Bonds dont on a déjà parlé en différentes circonstances. Euh, les... Τα project bonds λοιπόν, τι είναι, τίτλοι που εκδίδει μια εταιρεία που έχει δημιουργηθεί για αυτό το στόχο, για να χρηματοδοτηθούν έργα, ε, συγγνώμη, δραστηριότητες στον τομέα των ε, υποδομών ξέρετε ποιο είναι το rating το οποίο δίδεται. Οι χρηματοδότες προτιμούν τα 3α. Καμιά φορά και τα δύο. Προσπαθούμε λοιπόν να δούμε πώς οι τίτλοι που αφορούν κάποιο σχέδιο είναι, έχουν τέτοια εγγύηση, δίδουν τέτοια εγγύηση ώστε να προσελκύσουν τους επενδυτές με την συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάνουμε κάποιες προτάσεις. Δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες, αλλά κάθε φορά τι προσπαθούμε να κάνουμε. Προσπαθούμε να ε, αυξήσουμε τις πιστώσεις. Ίσως ε, χωρίζοντας το χρέος με τρόπο ώστε να το επομιστεί ένα μέρος του η ΕΤΕ και ένα μέρος οι άλλοι επενδυτέ. Εν πάση περιπτώσει δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, θα σας, εξηγώ ποιοι είναι οι τρόποι με του οποίου προσπαθούμε στα πλαίσια αυτή τη στρατηγική ε, για την Ευρώπη του 2020 να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προωθήσουμε τι δραστηριότητε μα. Μία δεύτερη παρατήρηση τώρα. Οι δραστηριότητε μα εντό Ευρωπαϊκή Ένωση θα επικεντρωθεί επίση στην καταπολέμηση τη κλιματική αλλαγή σας είπα προηγουμένως ότι το 2009 πέρσι υπογράψαμε δάνεια για σχέδια που αφορούν την μείωση των εκπομπών διοξιδίου συνολικού ύψους 17 δις και θα, θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση δεδομένου ότι το ΔΣ μας αποφάσισε ότι θα πρέπει προοδευτικά να αυξηθεί η αναλογία των δανείων μας προς αυτή την κατεύθυνση τα επόμενα χρόνια. Και προοδευτικά από 20% θα αυξήσουμε την, ε, τις δραστηριότητες μας σε αυτό το τομέα από ποσοστό 20% σε ποσοστό 25%. Συνοπτικά, κυρία Πρόεδρε, αυτές είναι οι δραστηριότητες μας εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά είμαι στη διάθεσή σας, εάν θέλετε, στις απαντήσεις που δώσω σε ερωτήσεις σας, σα μιλήσω για τις δραστηριότητες της ΕΤΕ και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβασή σα. Έχουμε έναν μακρύ κατάλογο συναδέλφων μου που θέλουν να σας κάνουν ερωτήσεις και θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ζητήσω συγγνώμη διότι θα πρέπει να παραστώ στις εργασίες μιας άλλης επιτροπής και θα δώσω την προεδρία στον συνάδελφό μου, τον κύριο Καρσία Μαργκάλιο. Και πάλι κύριε Μεστάτ σας ε, ε, ζητώ συγγνώμη, αλλά πρέπει να φύγω. La palabra ahora al señor Cutas. Το λόγο ζήτησε ο κύριος Κούτας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να καλωσορίσω και εγώ τον κύριο Μαϊστάτ που μας έδωσε τη δυνατότητα για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Να κάνω ένα προκαταρκτικό σχόλιο. Όλοι γνωρίζουν τη σημασία που έχει η τράπεζα του κύριου Μαϊστάτ στην Ευρώπη. Αναφερθήκατε επίσης και σε ποιους τομείς δραστηριοτήτων θέλετε να εμπλακείτε έρευνα και ανάπτυξη, αύξηση της δανειοδοτικής δραστηριότητας. Εδώ να μου επιτρέψετε να προσθέσω ένα στοιχείο. Να υπογραμμίσω την σημασία που έχουν τα κίνητρα για τις τοπικές οικονομικές δραστηριότητες και για τον ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι κυρίαρχο μέσο αυτό για την καταπολέμηση της ανεργίας, η οποία δυστυχώς είναι η πραγματικότητα σήμερα. Δεύτερον, σχετικά με τα λεγόμενα project bonds. Νομίζω ότι πρόκειται για μια καλή ιδέα. Όταν ξεκινήσετε με τα project bonds και όταν έχετε τη δυνατότητα να αναπτύξετε αυτή τη δραστηριότητα, σίγουρα θα βοηθήσετε πολύ στη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών. Πριν ε, έλθουμε εδώ, και ξεκινήσουμε τη συζήτηση αυτή, είχαμε συζητήσει τα θέματα των εγγυήσεων για τις ζημίες που προκαλούνται σε επενδυτικές δραστηριότητες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είπαμε ότι για να προστατεύσουμε και τα χρήματα των φορολογουμένων, είπαμε ότι η τράπεζά σας δεν θα πρέπει να αναλαμβάνει δραστηριότητες επενδυτικές σε χώρες οι οποίες χαρακτηρίζονται φορολογική παράδειση. Βέβαια τέθηκαν πολλές ερωτήσεις σχετικά με τους ορισμούς αυτών των χωρών. Δηλαδή τι είναι ένας φορολογικός παράδεισος σήμερα. Σαν εισηγητής για την ετήσια έκθεση ε, έχω ήδη επαφή Έχω ήδη έρθει σε επαφή και με άλλους συναδέλφους και με εκπροσώπους της τράπεζάς σας και νομίζω ότι κάποια πρώτα στοιχεία απάντησης τα έχουμε πάρει. Ευχαριστώ κύριε Κούτας. Και εγώ θα ήθελα να θέσω το θέμα των project bonds. Ο τρόπος με τον οποίο παρουσίασε ο κύριος Μπαρόζο ε, τα δείχνει με ένα πολύ ενδιαφέρον φως. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για τη βελτίωση των δικτύων τα οποία χρησιμοποιούμε και στον τομέα των μεταφορών και στον τομέα του περιβάλλοντος και στην ουσία αυτά είναι η σπονδυλική στήλη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Βέβαια όταν μπαίνει κάποιος σε λεπτομέρειες βλέπει ότι τα πράγματα είναι ιδιαίτερως περίπλοκα σε σχέση με τα project bonds. ο λόγος για τον οποίο μέχρι τώρα τα προγράμματα αυτά δεν έχουν προχωρήσει. Οι μονάδες αυτές ε, ε, δεν είναι έτοιμες, δεν είναι κερδοφόρες, δεν δίδει το κάθε κράτος τα απαιτούμενα ποσοστά ε, χρημάτων, δεν συνιστούν επιχειρηματική ευκαιρία. Τι ακριβώς συμβαίνει. Σίγουρα δεν αμφισβητώ τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να παρέμβει σε τέτοιου είδους προγράμματα, αλλά θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα για να καταλάβουμε καλύτερα. Έτσι ώστε αυτά τα project bonds να βοηθήσουν στην ολοκλήρωση του προγράμματος γιατί το θέμα αυτό ίσως τελικά μερικές φορές να συγχαίεται και με τη συζήτηση που γίνεται για τα ευρωομόλογα. Λοιπόν, τι θέλουμε. Θέλουμε ουσιαστικά να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό σε εισαγωγικά δημόσιο χρέος. Εάν ναι, ε, πώς αυτά τα project bonds θα πρέπει να επιστραφούν πώς θα πρέπει να αποσβεστεί η βάση περιπτώσει συγκεκριμένη δαπάνη ή επένδυση αν θέλετε. Είναι κάτι το οποίο θα συμπεριληφθεί στο χρέος σε το λεγόμενο εθνικό. Εν πάση περιπτώσει όλα αυτά είναι θέματα στα οποία θέλουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Υπάρχει επίσης και ένας φόβος εδώ διαφορετικός ότι η δημοκρατική νομιμοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων θα υπονομευθεί γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά ούτε και τα κοινοβούλια των κρατών μελών εμπλέκονται καθιοδήποτε τρόπο σε αυτές τις δραστηριότητες. Λάμπερτς. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ε, άκουσα ότι σίγουρα δεν είστε υποχρεωμένος να είστε ανάμεσά μας και εκτιμούμε γενικά την παρουσία σας ε, και σας ευχαριστούμε για αυτήν. Έχουμε ανάγκη από τον συγκεκριμένο αυτό διάλογο, ξέρουμε τον ρόλο που μπορεί να παίξει η τράπεζά σας και τι επενδυτικές δραστηριότητες υπάρχουν. Θα σταθώ και εγώ στο θέμα των project bonds. Δεν θα έλεγα ότι είστε πρόεδρε η τελευταία μας ελπίδα, αλλά είστε σαφέστατα ένα κομβικό ποσοστό σημαντικό της απάντησης που θα δώσουμε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Οι υψηλέ δανειοδοτικές σας δραστηριότητες σε τομείς όπως το, των, της μετρίασης των συνεπειών των κλιματολογικών αλλαγών είναι καλοδεχούμενες Παρόλα αυτά ε, η έλλειψη πιστώσεων στον τομέα αυτό θα ε, καταστεί ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα στο μέλλον. Ξέρετε ότι έχουμε προβλήματα και με κάποιες πρώτες ύλες όπως θα έχουμε σύντομα με το λίθιουμ και τα λοιπά. Ε, υπάρχουν προβλήματα για τα οποία και εσείς ε, προσπαθείτε να βοηθήσετε στη συνειδητοποίηση τους Πρέπει από τη μία να παρεμβαίνει κανείς σε κάποιους τομείς οι οποίοι είναι χρήσιμοι θα έλεγα, από την άλλη θα πρέπει να παρεμβαίνει όσο και λιγότερο μπορεί σε τομείς οι οποίοι είναι προβληματικοί διότι υπογόνοι κτλ. Τι κάνετε λοιπόν σε σχέση με προγράμματα τα οποία είναι βλαβερά για το περιβάλλον, για το κλίμα, για τις πρώτες ύλες, για το περιβάλλον γενικότερα έχετε μια σε εισαγωγικά θα χαρακτήριζα εσκεμμένη στρατηγική στον συγκεκριμένο τομέα γύρω από μια προοδευτική, από μια σταδιακή αποχώρησή σας, από μια αηφόρες ε, επενδυτικές δραστηριότητες. Ένα δεύτερο ερώτημα, να το εκφράσω αλλιώς, ε, βλέποντας ε, τα ποσοστά μέσα από τα οποία δραστηριοποιείστε, οι κανόνες της Βασιλείας, οι ρυθμίσεις της Βασιλείας που δεν έχουν περάσει στο νομικό μας πλαίσιο πλήρως ακόμα θα σας επηρεάσουν ή όχι. Ε, τα ποσοστά αυτά τα δέχεστε που προβλέπει η Βασιλεία 2 ή πιστεύετε ότι κάποιες από τις συστάσεις αυτές θα πρέπει να προσαρμοστούν στα ευρωπαϊκά δεδομένα για να αποφύγουμε στρεβλώσεις των πιστοτικών αγορών. Τώρα, τρίτη ερώτηση για την εξωτερική εντολή της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Καλείστε να παίξετε ένα ρόλο και εκτός συνόρων Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά γενική ομολογία δεν είσαστε σε επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης καταλήλως εξοπλισμένοι για τέτοιου είδους δραστηριότητες αναπτυξιακές. Συνεπώς ερώτηση τι κάνετε στο εσωτερικό της τράπεζας για να αυξήσετε τις εμπειρίες σας και την τεχνογνωσία η οποία απαιτείται για να αποφύγετε τα λάθη τα οποία έχουν κάνει διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και συνεχίζουν δυστυχώς να κάνουν στον τομέα τον επενδυτικό στην ανάπτυξη. Ευχαριστώ κύριε Λάμπερτς. Κύριε Μεστάτ έχετε το λόγο. Ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κούτας τον εισηγητή που με λεπτομεριακό τρόπο μελέτησε τις αστεριότητές μας. Για μας μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η ΜΜΕ είναι προτεραιότητα και τα δάνεια προς τις μεγάλες επιχειρήσεις θα μειωθούν, γιατί έχουν λιγότερο ανάγκη από τις ΜΜΕ. Και ξέρουμε ότι για τις ΜΜΕ παραμένουν οι δυσκολίες πρόσβασης στις πιστώσεις. Το διαπιστώνουμε και στην τελευταία μας έκθεση αυτό. Και βέβαια, ξέρω, ξέρουμε ότι οι μεγάλες τράπεζες υποβάλλουν σε περιορισμό στις ΜΜΕ που θέλουν να έχουν πρόσβαση σε επιστώσεις. Πέρσι, όπως σας είπα, ναι, ανήλθαν τα δάνειά μας σε 12 δις προς τις ΜΜΕ. Και σίγουρα και φέτος τα ίδια περίπου ποσά θα δανείσουμε. Και δανείζουμε τις τράπεζες υπό τον όρο ότι θα τις χρησιμοποιήσουν για να δανείσουν τις ΜΜΕ και οι συμβάσεις που ε, υπογράφουμε και οι όροι που μπορέσαμε εξαιτίας της κρίσης ε, να επιβάλλουμε στις ε, τράπεζες είναι κάτι που μας επιτρέπει να ελέγχουμε τον τρόπο με τον οποίο χορηγούνται. Και χαίρομαι διότι θα ασχοληθείτε εσείς ιδιαιτέρως με την καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων η πολιτική μας είναι η πιο αυστηρή σε τέτοιου είδους θέματα σε σχέση με τα άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Και γίνονται σε επίπεδο διεθνές ε, πολύ έντονη συζήτηση για αυτό το θέμα, διότι κάποιοι ε, εταίροι μας λέγουν ότι πάμε πολύ μακριά. Εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε πάρα πολύ αυστηροί και πρέπει να σας πω ότι είμαστε οι μόνοι οι οποίοι λέμε ότι θα πρέπει ε, ό,τι γίνεται να γίνεται στα πλαίσια κάποιων κανόνων όσον αφορά την ε, φορολόγηση. Και βεβαίως εμείς ακολουθούμε τους καταλόγους των ε, εξουσιοδιωτωμένων και επιστοποιημένων οργανισμών για τους φορολογικούς παραλύσεις. Ακολουθούμε τον κατάλογο της ΟΣΑ. Και στα πλαίσια της ομάδας ΓΚΑΦΗ που είναι η ομάδα που ασχολεί, εργασία που ασχολείται ε, για την καταπολέμηση του ξεπλήματος του βρώμικου χρήματος, ακολουθούμε κάποιους κανόνες, αλλά δυστυχώς ακολουθούμε τους κανόνες σύμφωνα με τους διεθνείς καταλόγους. Και μου λέγουν κάποιοι ότι δεν είναι πολύ σοβαρή αυτή η κατάλληλη Ίσως κάτι τέτοιο να συμβαίνει, αλλά αυτό είναι θέμα υποχρέωσης των κρατών μελών που είναι μέλη τέτοιων διεθνών οργανώσεων να αναθεωρήσουν αυτούς τους καταλόγους. Εμείς όμως δεν έχουμε την ικανότητα, την αρμοδιότητα, αν θέλετε, να καταρτήσουμε το δικό μας κατάλογο. Η κυρία Βόρτμαν έθεσε κάποιες πολύ εύστοχες ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, ποιοι είναι οι λόγοι της καθυστέρησης. Σωστά θέσατε το θέμα. Δεν είναι θέμα χρηματοδότησης ή καθυστέρηση, κυρίως στα πλαίσια των ε, ε, ευρωπαϊκών δικτύων. Υπάρχουν και άλλες δυσκολίες και καθυστερήσεις τεχνικής φύσεως, δυτικής φύσεως, έλλειψη συντονισμού ε, για την χορήγηση αδειών. Υπάρχουν πολύ σημαντικές καθυστερήσεις όσον αφορά τις απαλωτριώσεις πολλές φορές και πολύ, πολλές φορές μπορεί να είναι αντίθετη προς ένα έργο. Η καθυστέρηση για την ε, κατασκευή αυτών των διευρωπαϊκών δικτύων δεν είναι πάντα οφειλόμενες στη χρηματοδότηση. Τώρα, τα project bonds. Αυτό δεν είναι κάτι που ισχύει για οποιοδήποτε έργο υποδομής. Ισχύει μόνο για έργα υποδομής που θα έχουν επαρκή απόδοση για να μπορέσουν να προσελκύσουν και οι ιδιωτικού επενδυτές. Μίλησα για, χρηματοδο... για επενδυτές μαχροπρόθεσμα, δηλαδή όχι για κάποιον που θα απαιτήσει άμεση αποδόμπτηση, απόδοση. Η απόδοση μπορεί να προβλέπεται για αργότερα, αλλά θα πρέπει να είναι κατά κάποιο τρόπο σίγουρη. Όταν ένα συνταξιοδοτικό ταμείο επενδύει, δεν ζητά απόδοση ε, της επένδυσής του τον πρώτο χρόνο, αλλά πρέπει να είναι σίγουρο ότι σε 10-20 χρόνια θα είναι υπαρκή η απόδοση. Οι τίτλοι αυτοί εκδίδονται από ένα δημόσιο, από ένα συγγνώμη, ιδιωτικό φορέα. Δεν εξαρτώνται δηλαδή ούτε από τα κρατημέλη ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ιδιωτική εταιρεία η οποία εκδίδει τους τίτλους αυτούς και μπορείτε να φανταστείτε ότι έχει για τους, ε, το τμήμα senior, όπως λέγεται, για τους ιδιώτες και ένα τμήμα το οποίο αναλαμβάνουν η ΕΤΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, οι θεσμικοί επενδυτές μπορούν να είναι σίγουροι ότι θα έχουν απόδοση και θέλουν να επενδύσουν σε τέτοιου είδους σχέδια. Τώρα, από την μεριά της ΕΤΕ και του κοινοτικού προϋπολογισμού. Η επένδυση δεν θα είναι σημαντική απαραίτητο. Ο κίνδυνος όμως ε, είναι μεγαλύτερος για τον δημόσιο παρά για τον ιδιωτικό τομέα. Πρόκειται λοιπόν για τρόπους με τους οποίους προσπαθούμε να μειώσουμε το ρίσκο για τους ιδιωτικούς επενδυτές ώστε να τους προσελκύσουν αυτοί οι τίτλοι, πράγμα όμως που σημαίνει ότι ένα μέρος του κινδύνου το επομίζεται και το δημόσιο. δημόσιο τομέα. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άμεση επιπτώσεις για τις ε, δημόσιες επενδύσεις, γι' αυτό είπα ότι πρόκειται για κάποιο διαφορετικό για κάτι το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό από τα ευρωομόλογα. Τα project bonds λοιπόν είναι εντελώς διαφορετικά. Στα σχέδια των επόμενων χρηματοπιστωτικών προοπτικών μπορούμε να επέλεψουμε αυτό το θέμα, αλλά δεν πρόκειται περί αυτού του θέματος εδώ. Δεν έχουμε να κάνουμε με ευρωομόλογα. Ο κύριος Λάμπερτς μου έκανε μια ερώτηση για την τοποθέτησή μας σε σχέση με διάφορα σχέδια τα οποία δεν αφορούν, δεν είναι και τόσο ενδιαφέροντα όσον αφορά την μείωση των εκπομπών του Είναι σαφέ ότι όλο και περισσότερο τα σχέδια τα οποία χρηματοδοτούμε αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και είπαμε ότι το 20% για την παροή της ενέργειας θα πρέπει να αφορά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έχουμε ξεπεράσει αυτό το ποσοστό. Και πολλές φορές ακόμη χρειάζεται να χρηματοδοτήσουμε ε, εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν τον άνθρακα. Η Γερμανία, Φερρυπίν, έχει αυτό το περίφημο μίξ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως ξέρετε, έχει γίνει πολύ σημαντική προσπάθεια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά θεωρούν ότι ένα μέρος ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να παράγεται χρησιμοποιώντας τον άνθρακα. Και βεβαίως σε τέτοιους περιπτώσεις πρέπει να πληρούνται τρεις προϋποθέσεις. Να είναι σχέδιο αντικατάστασης. Δηλαδή να μπορέσει να αντικαστεί ένα μέρος της παραγωγικής ικανότητας. Δεύτερον, αυτό το νέο σχέδιο θα πρέπει να σημαίνει ότι θα υπάρχει μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος σε ποσοστό τουλάχιστον 20%. Και τρίτη κριτήριο πρέπει να είναι CCF ready. Δηλαδή το design αυτού του δέου εργοστασίου θα πρέπει να είναι έτσι γίνει όταν το, όταν το capture and storage project θα, μπορέσει να, θα είναι έτοιμο να μπορέσει να εφαρμοστεί από και να ακολουθηθεί από αυτό το εργοστάσιο. Δεδομένων λοιπόν των ιδιαιτεροτήτων της κάθε ε, εργοστασίου παραγωγής ε, ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα σχέδια. Ε, κατά την άποψή σας θα μειωθεί ή όχι παραγωγή σε αυτά τα πλαίσια. Μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι στην... για τη χρηματοδότηση της ε, ηλεκτρικής ενέργειας, όλο και περισσότερο στα διάφορα σχέδια που χρηματοδοτούμε, μειώνεται η αναλογία των στερεών καυσίμων. Αναφερθήκατε στην Συμφωνία Βασιλεία 3. Πιστεύουμε ότι κάποιοι κανόνες και στην πλαίσια της Βασιλείας 3, καθώς και αυτοί που ισχύουν ε, στα πλαίσια της International Accounting Board δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην πολιτική που ακολουθούν οι διάφορες εμπορικές τράπεζες στα πλαίσια του trading. Εμείς το ενεργητικό μας το διατηρούμε έως ότι έως ότου οριμάσει για να το διαθέσουμε. Το ενεργητικό μας, επαναλαμβάνω, εμείς το διατηρούμε μέχρι να οριμάσει ένα για να το διαθέσουμε. Υπάρχουν οι κανόνες της Βασιλείας 3 και κανόνες που συζητούν στα πλαίσια του Διεθνού Συμβουλίου Λογιστικών Προτύπων που δεν λαμβάνουν αρκετά υπόψη αυτή την ιδιαιτερότητα του μοντέλου δραστηριοτήτων που αναπτύσσουμε. Στείλαμε την προηγούμενη εβδομάδα στον Επίτροπο Μπαρνιέ ένα σημείωμα το οποίο προετοιμάσαμε με άλλα ε, ε, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και του ζητήσαμε να λάβει στο μέτρο του δυνατού υπόψη κάποιες τεχνικές συστάσεις τις οποίες κάνουμε. Και αν σας ενδιαφέρει αύριο το πρωί ε, το σεμινάριο του Eurofee οργανώνεται ένα σεμινάριο που αφορά τις ιδιαιτερότητες αυτές των μακροπρόθεσμων επενδυτών. Ευχαριστώ δεν απάντησα στο τελευταίο ερώτημα του κύριου Λάμπερτ, αλλά πρόκειται για μια συζήτηση που αν θέλετε μπορούμε να έχουμε κάποια άλλη φορά, δεδομένου ότι θα πρέπει να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Η ΕΤΕ μπορεί να παίξει το ρόλο μιας αναπτυξιακής τράπεζας και υπό συνθήκες. Αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο θα πρέπει να αποφασίσουν οι μέτοχοί μας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κάποια αμφισημία. Εάν η απάντηση είναι σαφώς ναι, καταφατική, θα πρέπει η ΕΤΕ και η ΕΤΕ θα πρέπει να παίξει το ρόλο αναπτυξιακής τράπεζας, θα πρέπει να αποδεχθούν όλοι ότι θα πρέπει να έχουμε τα μέσα. Ανθρώπινο δηματικό και όλα τα μέσα, τα τεχνικά και άλλα που χρειαζόμαστε, διότι εάν δεν μπορούμε να αποφασίσουμε με ποιο επιτόκιο θα πρέπει να δανείζουμε και τους φτωχούς δεν κάνουμε τίποτα. Έχουμε πάρα πολύ ε, το το κατάλογο συναδέλφοι θέλουν ερωτήσεις και αυτό παρακαλώ να είστε πάρα πολύ σύντομοι συνάδελφοι. Η Βίκη Φόρντ. κοιτάξτε, έχουμε ένα μακροσκελέστατο κατάλογο Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ όσοι υποβάλλουν ερωτήσεις για ένα μόνο λεπτό. Έχετε το λόγο, κυρία Φόρτ. Ε, κοιτάξτε, δεν απαντήσατε στην ερώτηση της κυρίας Βόρτμαν Κόλ σχετικά με την ε, δημοκρατική λογοδοσία. Ε, στο έγγραφο που μας στείλατε χθε ε, υπάρχει σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δαπανηθούν τα δημόσια κονδύλια από 1% μέχρι και 20%. Λέτε λοιπόν ότι αυτό δεν σημαίνει ότι αυξάνεται το χρέος των κρατομελών, αλλά επί της ουσίας αυξάνεται ο κίνδυνος με τον οποίο δαπανώνται τα δημόσια κονδύλια. Γιατί ενδεχομένως τα μετακινούμεθα σε μικρότερα ε, τμήματα, παρτίδες επενδύσεων ε, στον δημόσιο κυρίως ε, τομέα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει πραγματικά να κατανοήσουμε τον κίνδυνο που υπάρχει και να δούμε και την όλη υπόθεση από την άλλη πλευρά. Προφανώς στην Ευρώπη η υποδομή χρειάζεται χρηματοδότηση και τη χρειάζεται γιατί είναι πεπαλαιωμένη. Είτε πρόκειται για την ε, ενεργειακή ε, πρόκληση, είτε για την έρευνα και τις καινοτομίες. Όλα αυτά πρέπει να χρηματοδοτηθούν. Όμως, ακριβώς επειδή βρίσκεται σε κρίσιμη φάση η υποδομή, τα ΣΔΙΤ, ε, συμφωνώ με αυτά, τα ΣΔΙΤ αυτά έχουν και ηθικούς κινδύνους. Δηλαδή, τελικά ε, οι ιδιώτες ε, θα καθορίζουν το τι θα συμβαίνει στις επενδύσεις. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε περισσότερα κονδύλια και μεγαλύτερη λογοδοσία. Γι' αυτό και σας παραπέμπω ε, στην ερώτηση της κυρίας Βόρταν Κόλ που ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Και παρακαλώ να απαντήσετε. Καλημέρα κύριε Μεστάτ. Δίνω πολύ μεγάλη σημασία στην τράπεζά σας σαν μέσο αναπτυξιακό όχι μόνο της Ευρώπης αλλά και στο εξωτερικό και εγώ είμαι μέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης. Ε, να αναφερθώ σε μια λεπτομέρεια στην αναθεώρηση της εξωτερικής σας εντολής. Ε, μια υποσημείωση αναφέρεται η Ισλανδία σαν χώρα. Αν κατάλαβα καλά, οι επενδύσεις της ΜΠΕΗ στην Ισλανδία υπόκεινται σε κάποιες προϋποθέσεις προϋποθέσεις σε μια πιθανή συμφωνία για την επιστροφή ε, του χρέους που έχει η Ισλανδία προς την Ολλανδία και τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι αλήθεια κάτι τέτοιο, αν είναι αλήθεια είναι λυπηρό αυτό. Γιατί είναι μια μικρή χώρα και για μια τέτοια μικρή χώρα τέτοιου είδους λεπτομέρειες είναι απαράδεκτες. Δεν θα πρέπει να επιβραδύνονται οι επενδύσεις στην Ισλανδία γιατί η χώρα αυτή έχει ένα πρόβλημα με δύο χώρες μέλη. Κάτι τέτοιο δεν θα ήταν σωστό εν πάση περιπτώσει και δεν έχει σημασία και δεν θα διευκολύνει την επιστροφή του χρέους της Ισλανδίας προς τις δύο αυτές χώρες. Μπορείτε να μου δώσετε κάποιες λεπτομέρειες. Ευχαριστώ κύριε Μπέρναρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να επανέλθω ε, σε αυτό το θέμα των ε, καινοτόμων εργαλείων χρηματοδότησης. Αναφερθήκατε και εσείς σε αυτά σήμερα το πρωί και η Κομισιόν παλαιότερες και νύν αναφέρονται τις τελευταίες εβδομάδες σε ομόλογα στην μόχλευση του κοινοτικού προϋπολογισμού. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά καινοτόμα εργαλεία και θα μου άρεσε εξήγηση. Θα ήθελα όμως και να δω πού ακριβώς βρισκόμαστε όσον αφορά την διαχείριση κινδύνων. Αναφέρατε ότι η τράπεζά σας θα αναδιαρθρώσει ε, τα χρέη, θα τα ανασυστήσει. Ε, ορισμένες τράπεζες το κάνουν αυτό τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν ε, βεβαίως επικρίνουμε τις ε, τράπεζες εδώ στο Κοινοβούλιο για αυτά τα οποία κάνουν στις αναδιαρθρώσεις. Πρέπει να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια οποτεδήποτε χρησιμοποιούνται τέτοια είδους εργαλεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτον, ποιο θα καθορίζει τη μόχλευση, το επίπεδο μόχλευσης. Δεύτερον, υπάρχει, υπάρχουν εμπειρογνώμονες και ποια είναι η πολιτική σε σχέση με τα ειδικά εργαλεία και τελικά ε, ποιος ε, συμβουλεύει, ποιες τράπεζες συμβουλεύουν την ε, τράπεζα επενδύσεων για τέτοιου είδους καινοτόμα θέματα. Ο κύριος, η κυρία Στήλα Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και κύριε Μαϊστάτε για την ε, παρέμβασή σας. Εγώ πρέπει να σας πω συμφωνώ με πολλά αυτά που ελέγχθησαν. Ε, όσον αφορά την προοπτική των ΜΜΕ, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συμφωνώ μαζί σας που είπατε ότι εξακολουθεί να υπάρχει ένα πρόβλημα με τη χρηματοδότηση αυτών. Ε, θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε πώς μπορούμε να βρούμε λύση σε αυτό το πρόβλημα. Γιατί νομίζω το 92% είναι οι μικρομεσαίες των επιχειρήσεων μας. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπους να τις βοηθήσουμε, ε, όχι μόνο μέσα από ε, επενδύσει σε μεγάλε εταιρείε, όπω είπατε, αλλά να δώσουμε προτεραιότητα στις μικρομεσαίες. Ε, θα ήθελα την προοπτική της έρευνας και να μας πείτε πώς ακριβώς μπορούμε να αμβλύνουμε κινδύνους και αυτό το στοιχείο να τη συμπεριλάβουμε στην Ατζέντα 2020. Ίσως μπορείτε να αναφερθείτε συγκεκριμένα σε προγράμματα. Μιλάμε για την ψηφιακή Ατζέντα. Ε, γιατί ακριβώς σε πράγμα μιλάμε. Θα ήθελα να έχω λεπτομέρειες από αυτού. Και ένα άλλο θέμα ε, που θα ήθελαν και άλλοι συνάδελφοι να ενημερωθούν, τα project bonds, τα περίφημα. Πολλοί στις εκλογικές μας περιφέρειες ε, έχουμε προγράμματα υποδομής. Αυτή τη στιγμή υπάρχει έλλειψη χρηματοδότησης, τουλάχιστον στη δική μου την εκλογική περιφέρεια. Αυτά λοιπόν τα project bonds είναι πολύ ενδιαφέροντα. Ε, μας ενδιαφέρει και θέλουμε περισσότερες ε, πληροφορίες. Ε, είναι ένα σημαντικό εργαλείο και πρέπει να εξεταστεί. Σας ευχαριστούμε για αυτά που είπατε σήμερα το πρωί. Λυπάμαι που δεν υπάρχουν και άλλα μέλη εδώ, γιατί αυτά που κάνετε είναι πολύ ενδιαφέροντα για μας και πραγματικά πρέπει να τα στηρίξουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Τατή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αναφέρατε μεγάλα σχέδια υποδομών, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, τεχνικά προβλήματα, χρηματοπιστωτικά. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση για μια μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη, κάπως σε πιο ανθρώπινο επίπεδο. Ίσως μικρότερης εμβέλειας από ό,τι αναφέρατε κατά τη διάρκεια της παρεμβασής σας και από ό,τι είπαν οι συνάδελφοι. Τι μπορεί να κάνετε για να μπορέσει να βοηθήσει τους νέους να καταπολεμήσουν την ανεργία και να ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας. Σήμερα το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των νέων 14-25 είναι της τάξεως του 20%, στην Ισπανία του 24%. Νομίζω ότι μπορείτε να διαδραματίσετε κάποιο ρόλο. Τις επόμενες εβδομάδες θα οργανωθεί ένα συνέδριο στο Παρίσι για τα θέματα απασχόλησης που αφορούν τους νέους. Θα έχουμε ανάγκη και από την ε, δική σας συνδρομή και πρέπει να σας πω ότι τις 15 Σεπτεμβρίου έθεσε σε κίνηση ένα πρόγραμμα η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, που αφορά τους νέους εγκινήσεις στην Ευρώπη. Πρέπει να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μελετά τη δυνατότητα να σε σε συντονισμό με την ΕΤΕ δάνεια για τους νέους για να μπορέσουν να μετακινούνται στην Ευρώπη να σπουδάζουν και μπορέσουν να ενταχθούν στην ε, αγορά εργασίας. Το 2011 θα έχουμε κάποια αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας. Μπορείτε να μας πείτε εσείς τι κάνετε σε αυτό το τομέα, διότι πιστεύουμε ότι θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε. Είναι κάτι το οποίο επιθυμούμε και θα θέλουμε να μας πείτε εσείς πώς μπορείτε να κάνετε κάτι τέτοιο. Ο κύριος Φρέιρε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις εξηγήσεις που μας δώσατε για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα project bonds. Και να ρωτήσω το εξή. Μας εξηγήσατε ότι τα project bonds θα έχουν σχέση με την μεγάλα σχέδια που αφορούν τα έργα υποδομής και με την λειτουργία και ιδιωτικών ε, σχεδίων. Υπάρχουν χώρες που δεν έχουν προβλήματα με τον υποδοτών, αλλά έχουν τεχνικά προβλήματα ή τεχνολογικά. Θα μπορούσαν τα project bonds να εφαρμοστούν ε, σε τέτοιου, για τέτοιου είδους θέματα στα πλαίσια της στρατηγικής του 2020 και θα μπορούσαν ενδεχομένως τα project bonds να αντικαταστήσουν ε, κάποιες χρηματοδοτήσεις που καθόρισε η τράπεζα. Δηλαδή δάνεια που αφορούν ε, σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας, όπως στην περίπτωση Πορτογαλίας και Ισπανίας. Πιστεύω ότι υπάρχει μια δέσμευση προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτά τα project bonds θα μπορούσαν να ε, συμπληρώσουν τέτοιου είδους ε, δάνεια είναι να τα αντικαταστήσουν. Ευχαριστώ κύριε Τσικλώνα. η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, μπορεί να εκπονεί κανόνε ε, για πολύ σημαντικά δάνεια στα κράτη-μέλη και υπάρχουν και πάρα πολλοί ανταγωνιστέ. Όταν λοιπόν επειδή τελικά ένας κερδίζει τον ε, διαγωνισμό, όταν διαπιστώνονται ανομαλίες που μερικές φορές ευσταθούν κιόλας, Ποιο είναι ο δικό σα ο ρόλο, Εσεί κάνετε έρευνε. Αναλαμβάνετε το ρόλο της Όλαφ. Ευχαριστώ κύριο Σβέγγλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δώσατε το λόγο. Ε, έχω μία ερώτηση για αυτό που είπε ο κύριος ε, Μάιστατ. Πρώτον, κατάλαβα καλά ότι μπορείτε να έχετε τα στοιχεία εκείνα που δείχνουν τη χρηματοδότηση σε πράσινους τομείς σε αντίθεση με τη χρηματοδότηση σε παραδοσιακούς ε, τομείς ε, όπου εξακολουθεί να γίνεται εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών ε, και της μη ανακυκλώσιμης ενέργειας. Έχετε τέτοιου είδους στοιχεία. Και δεύτερον, εγώ δεν ήξερα ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συμμετέχει στην χρηματοδότηση ε, εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, μίγματος ενέργειας στη Γερμανία. Μήπως μπορείτε να μας πείτε το πώς ακριβώς χρηματοδοτούνται τα, ε, οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από άνθρακα στη Γερμανία. Μήπως μπορείτε να τοποθετηθείτε επ' αυτού. Παρακαλώ, έχει το λόγο. Γνωρίζουμε ε, για τον λίγο χρόνο που υπάρχει. Εν πάση θα απαντήσω τηλεγραφικά. υπήρξαν ε, πολλές ερωτήσεις σχετικά με τα project bonds. Έχουν προκαλέσει ενδιαφέρον, είναι κάτι το καινοτόμο. Λογικό είναι. Εμείς δεν μπορούμε να προσφύγουμε στην τεχνική αυτή για, οποιοδήποτε, για οποιαδήποτε επένδυση. Μιλάμε μόνο για επενδύσεις, για σχέδια, για προγράμματα που έχουν μια διασφαλισμένη αποδοτικότητα σε δεδομένο χρονικό διάστημα και υπάρχουν κάποιε μορφές υποδομών που δεν προσφέρονται προς την κατεύθυνση αυτή. Πρόκειται για προγράμματα πολύ σημαντικά για την περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά δεν δίδουν σε καμία περίπτωση εγγυήσει ε, στου εργολάβου θα έλεγα, σε αυτούς που τα προωθούν και τα κατασκευάζουν επαρκή έσοδα εγκαίρως. Πρόκειται λοιπόν για κάποια προγράμματα για τα οποία ο χρήστης άμεσα πληρώνει και βοηθά στην απόσβεση της επένδυσης για τον σε εισαγωγικά ε, επιχειρηματία. Θα τα συζητήσουμε αυτά λεπτομερέστερα. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα στη συγκεκριμένη περίπτωση μεγαλύτερης δημοκρατικής νομιμοποίησης από ότι σε άλλες οικονομικές ή χρηματοπιστωτικές παρεμβάσεις. Όταν χρησιμοποιούνται τα δημόσια χρήματα και στη δραστηριότητα αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει τις ίδιες αρμοδιότητες που έχει και ε, ε, ε, στα υπόλοιπα χρηματοδοτικά μέσα. την κοινή Στήλερ. Θα ήθελα να πω ότι όλα τα προγράμματα τα οποία θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε στα πλαίσια της στρατηγικής Ευρώπη του 20 δεν μπορεί να χρησιμοποιήσουμε μόνο τα project bonds. Είναι ένα μέσο ανάμεσα σε άλλα τα project bonds. Υπάρχει και άλλο ένα μέσο το οποίο υπάρχει, είναι ε, το χρηματοδοτικό μέσο ανακατανομής, το Resharing Finance Facility. Αυτά είχαν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα για ερευνητικά, στο ερευνητικό πεδίο μόνο. Έχουμε τώρα μία έκθεση ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων που έχει ε, εκτιμήσει αυτό το σχέδιο και θεωρεί ότι η χρήση του μέχρι τώρα ήταν σχετικά θετική και θα πρέπει το σχέδιο αυτό, το Resharing Finance Facility, να χρησιμοποιηθεί και περισσότερο και να καλύψει ό,τι έχει σχέση με την καινοτομία. Να διευρυνθεί δηλαδή η ε, χρήση του και σε τομείς όπως η ψηφιακή ατζέντα σαν παράδειγμα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ε, το μέσο αυτό στο σύνολο των καινοτομικών δραστηριοτήτων συσταγωγικά. Για τον κύριο Μπέρμαν. Θα διαπιστώσω ότι το Συμβούλιο ε, προσέφεσε την υποσημείωση αυτή για την Ισλανδία μετά από αίτημα δύο χωρών. Εγώ δεν πήρα μέρος στις συζητήσεις αυτές και δεν το πρότεινα. Για την κυρία Ντατή. Έχω την αίσθηση ότι υπογραμμίζεται ένα πρόβλημα το οποίο αποκτά σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δραματική διάσταση. Δεν είμαι σίγουρος όμως ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι το κατάλληλο μέσο για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ανεργίας των νέων. Λόγω ακριβώς του καθεστώτος μας δεν μπορούμε παρά να χρηματοδοτούμε επενδυτικές παρεμβάσεις και δραστηριότητες. Επεκτείνουμε θα έλεγα τον ορισμό των επενδύσεων ακόμα και σε επίπεδο άειλων εισαγωγικά επενδύσεων αλλά δεν μπορούμε να παρέμβουμε παντού. Εφόσον υπάρχουν επενδύσεις η τράπεζά μου θα παρεμβαίνει εκεί μόνο. Στον κύριο Σικλούνα. Πράγματι αυτό είναι τμήμα της δραστηριότητάς μας. Όταν χρηματοδοτούμε κάτι βλέπουμε αν ο επιχειρηματίας σέβεται τους ευρωπαϊκούς κανόνες σε ό,τι έχει σχέση με τις προμήθειες, ε, τους διαγωνισμούς και τους περιβαλλοντικούς κανόνες. Αυτοί είναι οι δύο τομείς άλλωστε που δίνουν ε, θα έλεγα ευκαιρίες για περαιτέρω επαφές με τους ε, οικονομικούς εμπλεκομένους. Εμείς ε, δεν ξοδεύουμε τα χρήματά μας άμα δεν είμαστε βέβαιοι για τον σεβασμό των κανόνων των δημοσίων προμηθειών και του σεβασμού του περιβάλλοντος. Για τον κύριο Γκίγκολντ, σχετικά τώρα με τα ποσοστά, ποιο είναι το τμήμα των ε, μονάδων παραγωγής που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα. Θα σας δώσω τις λεπτομέρειες αυτές σε συγκεκριμένα παραδείγματα χρηματοδότησης της τράπεζάς μας κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι σεβαστήκατε το χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Σας ευχαριστώ και για την ευκρίνεια των θέσεών σας. Vamos a proceder Η ψηφοφορία. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ζητήσω από τις κυρίες και τους κυρίους ε, συναδέλφους να δοκιμάσουν τις ε, κάρτες τους για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. va voter. test n'est Λοιπόν, δεν κάνατε ακόμη το τεστ, έτσι. ¿Dónde se vota May you vote, please. για το τεστ, παρακαλώ. Todavía tienen que chequear porque están lejos de 35, 34. ¿Qué pasa? Eh, que no todos han verificado, pero bueno. We have only 31 and we should be 38. That's... 31 μόνο ψήφισαν και πρέπει να είμαστε 38. Για ψηφίστε παρακαλώ όλοι. A vote. I know, I know. Ahora sí. Ah, hay, un, hay uno más de los socialistas. Tienen que quitarlo. Okay, now the, we have a problem with the socialist group. We have what... Έχουμε ένα πρόβλημα με τη σοσιαλιστική ομάδα. Έχουμε έναν περισσότερο από ό,τι πρέπει. Too much. now it's okay. Okay. Okay, there we go. So we have two persons from the PP who have... Τι συμβαίνει, κάποιος από το Έλκο, ο κύριος Κάζας και η κυρία Λούλιν δεν έχουν κάρτες. Λοιπόν, ψηφίζουμε πρώτα απ' όλα για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Συντάκτρια γνωμοδότησης η κυρία Πιετικάινεν, τροπολογία 15, Αντολίν, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 16 του ιδίου, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δύο της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία, παράγραφος 2 του άρθρου 3. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 17. Σάντσες Πρεσέδο. Συγγνώμη, πάμε στο 20. Στην... Περνάμε την 20 του κυρίου Κανφίν. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 Σμιτ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 άρθρο 4 Ashley Fox. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28. Όχι. Ναι, 28 λέει πάλι ο πρόεδρος. Φόξ, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 29, Σμιτ, υπέρ, κατά. Η ηλεκτρονική επαλήθευση. Τροπολογία 29. Έληξε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 22 προς 18. 30 Φόξ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. εγκρίνεται με 21 προς 18. Συμβιβαστική τροπολογία για την νέα παραγραφο 3 του άρθρου 5. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 32. Παρεμφερεί με την 33. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 34. Φόξ, υπέρ. Χωρίς τι ψηφοφορία που ζήτησε η συγγήτρια. Το πρώτο μέρος φτάνει μέχρι ψηφίζ... μέχρι το κείμενο το οποίο τροπολογήθηκε το έτσι όπως προβλέπουν τα άρθρα 9, 11, 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος, το υπόλοιπο μέρος του άρθρου υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 35. Σμιτ. Θέλετε ηλεκτρονική παρήθευση. Εντάξει, για το δεύτερο μέρος. Έληξη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Έκανα λάθος, λέει ο πρόεδρος. 35. Σμιτ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 35. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 22 προς 17. 36. Φοξ για διαγραφή. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 37. Χωριστή ψηφοφορία. Το πρώτο μέρος αφορά τα σημεία α έως και γ. Υπέρ, κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται το πρώτο μέρος. Περνούμε στο δεύτερο, το σημείο δέλτα. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 39 Φόξ για διαγραφή. Υπέρ. Κατά. Αποχή ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει ψηφοφορία. Ναι, στην 39, την 39 ψηφίζουμε. Όχι, λέει ο πρόεδρο. Την 38 ψηφίζουμε. Okay. sorry. Συγγνώμη, λέει ο πρόεδρο. Την 38 ψηφίζουμε. Ξαναρχίζουμε. Ξαναρχίζουμε για την 38. Για διαγραφή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 39. Επίσης για διαγραφή. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Εγκρίνεται. Με μεγάλη πλειοψηφία. 40. Fox. Άρθρο 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 41. Fox. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 42 Fox. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 43 για διαγραφή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 44 Ναι, ναι, διαγράφεται η, η, η παράγραφος. Εγκρίθηκε 43. 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 46 φόξ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση τη 46. Αρχίζει ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 47. Καμφά. Υπάρχει μία προφορική τροπολογία του άρθρου 20. Υπέρ. Υπάρχει προφορική τροπολογία, επαναλαμβάνει ο πρόεδρος στα γαλλικά, στην τροπολογία 47. Γίνεται κάποια παρατήρηση χωρίς μικρόφωνο από την αίθουσα. On a des problèmes. Okay. If the oral amendment is adopted, the original text falls. So we are voting on the on the oral amendment. Ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία υπέρ. Όχι. Από... Ακούστε, ας κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Τι ψηφίζουμε, πρόεδρε, ρωτάει κάποιος. ποια ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε την ε, προφορική τροπολογία του 47. εγκρίνεται, άρα καταπίπτει η 47. 48 καμφά. Πρώτα απ' όλα ψηφίζουμε και εδώ την προφορική τροπολογία. Υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία για την προφορική τροπολογία. Λίγη ψηφοφορία. εγκρίνεται. Προς 22 προς 21. Luego son 23 votos a 21. De acuerdo, la enmienda 40. Καταπίπτει 48 λοιπόν και 49. Υπάρχει τρομερή σύγχυση. Μπορούμε να κάνουμε πάλι μια επαλήθευση. Διότι υπήρχε τρομερή σύγχυση. Δεν ξέραμε τι ψηφίζαμε. Λοιπόν, τροπολογία 48. Του άρθρου 20, παράγραφος 3. Αρχίζει η ψηφοφορία. Και πάλι λέει ο πρόεδρος. Λίγη ψηφοφορία. συμπεριλαμβανομένης και της κυρίας Κράτσα 24-19. Θα ψηφίσουμε τώρα την ε, τροπολογία 49 ε, καταπίπτει. Ψηφίζουμε την 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 51 Fox υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 52 Fox υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53 Fox για διαγραφή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 φόξ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 55 υπέρ κατά αποχές Ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει ψηφοφορία. Τις 55. Λίγη ψηφοφορία. 24 προς 20. Εγκρίνεται. 56 Fox υπέρ. Κατά. Αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση της 56. 30 προς 13 εγκρίνεται. 57. Σμιθ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 58. Φόξ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. 29 προς 13 εγκρίνεται. 59 Fox. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 60 Fox υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61 Fox υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 Σμιτ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 64 κονφά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 65 κονφά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 45. Συμβιβαστική τροπολογία. Για το άρθρο 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει η 67 και πάμε στις Τελική σκέψη. Σαρή Εσάγια, 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 4 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται, 11 συμβαστική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 6 Συγγνώμη, 7, 7 τη εισηγήτριας, διορθώνει ο πρόεδρος. Υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. 25 προς 19 εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία για την 11α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 νέο, 8 όλες σμιτ υπέρ κατά εγκρίνεται. Στο 12 υπάρχει προφορική τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 39. Εάν εγκριθεί, καταπίπτει η 12 Σμιτ, υπέρ της προφορικής τροπολογίας υπέρ. Για να παρακαλέσω όλους τους χριστιανοδημοκράτες να ψηφίσουν. Προφορική τροπολογία της αιτιολογικής σκέψης 39 επαναλαμβάνει πρόεδρος. Προφορική τροπολογία. θα ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία του 39, λέει ο Πρόεδρος. Βουζαβέ. αυτός είναι ο κατάλληλος του Πρόεδρου. Αιτιολογική σκέψη 39. Αν ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία, η 12 καταπίπτει. Θα ψηφίσουμε πρώτα την προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρα δεν θα ψηφίσουμε τη 12. Πάμε με τον ίδιο τρόπο να ψηφίσουμε την Προφορική τροπολογία που αφορά την ιδεολογία 57. Υπέρ, κατά. Εγκρίνεται, άρα δεν ψηφίζουμε τη 13. Στην 60. Παρακαλώ. Θέλω να παρατηρήσω, Πρόεδρο, ότι ίσως ο κατάλογος ψηφοφοριών έχει γίνει με τρόπο ώστε δεν ψηφίσαμε την προφορική τροπολογία του κυρίου Σμιτ, αλλά τη εισηγήτριας. Και μετά έχουμε την ψηφοφορία του Σμιτ. Εγώ δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο. Άκουζαν Πολ. Εάν ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία, δεν θα ψηφίσουμε την τροπολογία Σμιτ. Η προφορική τροπολογία δεν αφορά την τροπολογία Σμιτ, άρα τη συζυγήτρια τροπολογία. Από τη στιγμή που το ψηφίσαμε, το υπόλοιπο κομμάτι καταπίπτει. Considerando 69, enmienda 1. Λοιπόν, η τελική σκέψη 60 καινούρια. Τροπολογία είναι τη εισηγήτριας. Υπέρ, κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Εγκρίνεται. Άρα Καταπίπτει η 14. Ψηφίζουμε το κείμενο έτσι όπως το τροποποιήσαμε. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. 38 υπέρ και 3 κατά. Και ψηφίζουμε το ψήφισμα το νομοθετικό ψήφισμα. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει, λίγη. Λίγη ψηφοφορία. 36 προς 3 εισηγήτρια, σας συγχαίρουμε. Προχωρούμε. Διασφάλιση ανεξάρτητων εκτιμήσεων επιπτώσεων. Συντάκτης γνωμοδότης ο κύριος Επινγκ. Λοιπόν, τελείωσε το διάλειμμα. Ψηφίζουμε. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση αρχίζει ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. 22 προς 17. Εγκρίνεται. Παράγραφος 2. Το αρχικό κείμενο. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 4. Τροπολογία μαν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. 20 προς 20 λέει ο πρόεδρος. Ο κύριος Μαν. Εγώ πήρα μέρος και στην προηγούμενη ψηφοφορία. Μέχρι τώρα δεν είχα την κάρτα, αλλά από εδώ και πέρα και μιας και η κυρία Κράτσα δεν είχε ψηφίσει ακόμα, θεώρησα ότι δεν ήταν απαραίτητο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πήρα μέρος στην τελευταία ψηφοφορία να με καταγράψετε. 22-20 είναι το αποτέλεσμα, συνεπώς. Η ελληνογερμανική συνεργασία θριάμβευσε. Ήταν 22 a 20 en Άρα είχαμε το, ε, έγκριση με 22 προς 10. Παράγραφ, παράγραφος 4, τροπολογία 4, Mann. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Της τροπολογίας 4. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. 21-19. Αποφασίζουν ε, αυτοί που δεν έχουν κάρτα. Συνεργασία ελληνογερμανική. Δουλεύει το σύστημα. Παράγραφος 5. Χωριστή ψηφοφορία. Το, όλο το κείμενο χωρίς τις λέξεις, όχι σε περιπτώσεις, μέχρι διαδικασία συναπόφασης. Οι σοσιαλιστές ζήτησαν χωριστή ψηφοφορία. Ναι, ναι, ζήτησαν οι σοσιαλιστές χωριστή ψηφοφορία, λέει ο πρόεδρος, απαντώντας σε κάποιους συναδέλφους του, του οποίου δεν ακούμε, διότι μιλούν χωρί μικρόφωνο από την αίθουσα. Ο δικός μου κατάλογος ψηφοφοριών λέει το εξής. Θα ψηφίσουμε το πρώτο τμήμα εκτός από τη φράση που λέει εκτός από τις περιπτώσεις. Ε, αυτό είπα λέει ο Πρόεδρος. Θα ψηφίσουμε το κείμενο χωρίς αυτό το τμήμα. Αυτό είναι το πρώτη, η πρώτη ψηφοφορία και η δεύτερη ψηφοφορία θα είναι οι υπόλοιπε λέξεις. Μα αυτό είπα λέει ο Πρόεδρος. Χωριστή ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε πρώτα απ' όλα όπως είπα και προηγουμένως, το κείμενο, χωρίς τις λέξεις, μόριο της φράσης που αρχίζει με only και τελειώνει με procedure. Αυτό είπα και εγώ. Έτσι λοιπόν, επαναλαμβάνω, ψηφίζουμε χωρίς αυτές τις, αυτό το ε, κομμάτι της πρότασης. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε αυτό το κομμάτι της φράσης. Υπέρ, κατά, αποχές, ε, ηλεκτρονική επαλήθευση. Λίγη η ψηφοφορία. 21 προς 19 υπέρ. Λοιπόν, τη σκέψη Α. Τροπολογία 1 Τόμας Μαν. Εγκρίνεται. Στο Β. Τροπολογία 2 του κυρίου Μαν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Λίγη ψηφοφορία. 24-16. Εγκρίνεται. Γάμα. Το πρωτότυπο κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. 21 προς 20. Δέλτα. Το πρωτότυπο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το κείμενο έτσι όπως τροπολογήθηκε. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. 29 προς 11 Συγχαίρω τον εισηγητή. Το επόμενο θέμα De acuerdo, vamos a votar. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε την επανεξέταση των κανόνων για τις συμφωνίες οριζόντιας συνεργασίας. Πρόκειται για ερώτηση για προφορική απάντηση. Πρόκειται για το σημείο 14 της ημερησίας διάταξης. Είμαστε έτοιμοι. Ε, στο εισαγωγικό μέρος, τροπολογία 1 σουάμπ. Υπέρ κατά εγκρίνεται. 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 των σοσιαλιστών. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 των σοσιαλιστών. Υπέρ. Όχι, όχι, όχι. Συγγνώμη. Συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Στην παράγραφο 2 ψηφίζουμε το πρωτότυπο. Υπέρ Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Παράγραφος 3. Τροπολογία 4 των σοσιαλιστών. Υπέρ, κατά, ε, αποχές. Το πρωτότυπο εγκρίνεται. Παράγραφος 5. Το πρωτότυπε. Σουάμπ. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το κείμενο έτσι όπως το τροποποιήσαμε με ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχή Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. 40 υπέρ. Εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στην πρόταση νομοθετικού ψηφίσματος που συνοδεύει αυτή την προφορική ερώτηση. Παράγραφος 1. Τροπολογία 1 των σοσιαλιστών. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2. Τροπολογία 2. Με προφορική ερώτηση από το Call on the Commission και τα λοιπά και τα λοιπά μέχρι το Stakeholders. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. τρία των σοσιαλιστών. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. τέσσερα... Πρωτότυπο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 5. Πρωτότυπο υπέρ κατά εγκρίνεται. Παράγραφος 6. Το πρωτότυπο υπέρ κατά εγκρίνεται. Παράγραφος 7. Τροπολογία 4 σοσιαλιστών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 σοσιαλιστών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 9. Τροπολογία 6 των σοσιαλιστών πρωτότυπο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 στην παράγραφο 10 των σοσιαλιστών. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10. Φιλίπ Λαμπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Πρωτότυπο. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 του κυρίου Λαμπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 12. Με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος. Τροπολογία 12 των σοσιαλιστών. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Λίγη ψηφοφορία. 20 προς 21 απορρίπτεται. Όχι, 18 προς 23. Απορρίπτεται, λέει ο Πρόεδρος. Ψηφίζουμε το πρωτότυπο. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 14. 13, τροπολογία 13 του κυρίου Λομπέρ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Στην παράγραφο 15 ψηφίζουμε το πρωτότυπο κείμενο. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις α έως δ εγκρίνεται. και το πρωτότυπο citation 1 με 13 εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το κείμενο έτσι όπως τροποποιήθηκε με ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη η ψηφοφορία. 38 πλειοψηφία. Εγκρίνεται λοιπόν απόλυτη και τελειώσαμε με τις ψηφοφορίες. Και περνούμε στο επόμενο θέμα terminado el... Uh, uh, Hello, Peter. Terminado el voto, pasamos ahora a discutir... Λοιπόν, τελειώσαμε με την ψηφοφορία και θα συζητήσουμε τώρα την έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2009. Εισηγητής ο κύριος Έπινγκ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η πολιτική ανταγωνισμού είναι η ε, πολιτική πυρήνα της ε, Επιτροπής γιατί καθιστά την Επιτροπή ισχυρή. Όμω, ποιο είναι αρμόδιο για αυτή την πολιτική. Ο κύριος Μάντελσεν, επίτροπο εμπορίου, γράφει στο βιβλίο του με επικεφαλίδα Τρίτο άνθρωπο και παραθέτω. Από τη στιγμή που είχα ξεκινήσει την ε, καθημερινότητά μου, το βασικότερο εμπόδιο που έπρεπε να ξεπεράσω ήταν να είμαι ε, το αφεντικό του σπιτιού μου, σε εισαγωγικά. Δυστυχώ ο κύριο Κίνερ δεν είναι εδώ. Όπω όλοι ξέρετε, ο κύριο Μάντελσεν είναι ο άνθρωπο παντό καιρού και παρόλα αυτά όμω δεν τα κατάφερε. Ε, τώρα αυτή η επιτροπή είναι υπό τον κύριο Αλμούνια. Ο κύριος Αλμούνια είναι άραγε κύριος ε, και αφεντικό του τομέα του. Πέρυσι συμφώνησε με την έκθεση Ινεφέλτ, πράγματι δεν χρειάζεται να επανανακαλύψουμε τον τροχό. Το ερώτημα που τίθεται είναι τι θα κάνουμε στο μέλλον. Υπάρχουν λοιπόν δύο-τρία θέματα που θέλω να προσθέσω. Πρώτον, όσον αφορά τι κρατικέ ενισχύσει. Η Κομισιόν θέσπισε προσωρινού κανόνε για να αντιμετωπιστεί η κρίση. Όμω, ε, είναι αυτό που λέμε ουδέν μονιμότερον του προσωρινού μήπως πρόκειται περί αυτού. Άρα δηλαδή χρειαζόμαστε μεγαλύτερες ε, διευκρινήσεις για το θέμα του phasing out. Δεύτερον, ο στόχος της πολιτικής ανταγωνισμού είναι να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού που διασφαλίζουν τον θεμητό ανταγωνισμό που είναι υποφελής για τους καταναλωτές, τουλάχιστον αυτή, αυτό είναι το νήμα της σκέψης. Κατά τη διάρκεια της κρίσης άλλαξαν τα πράγματα. Σε ορισμένε περιπτώσεις η Κομισιόν χρησιμοποίησε αυτή την πολιτική ως δούριο ύπο για να αναδιαρθρώσει ένα ολόκληρο τομέα. Κυρίως τα κριτήρια για τι επενδύσεις ε, και τις κρατικές ενισχύσεις ήταν ασαφή. Ε, μάλιστα η Κομισιόν ε, περιόρισε, σμίκνε τις επιχειρήσεις και έτσι μετέτρεψε Ευρωπαίους παγκόσμιους παίκτες σε περιφερειακούς παίκτες και συνέβη και το αντίθετο. Δέστε παραδείγματος χάρη την ΚΑΜΠΕΣΕ η ευρωπαϊκή οικονομία, κύριε Πρόεδρε, χρειάζεται ανταγωνιστικού παίκτε στην παγκόσμια αγορά για να μπορεί να ανταγωνιστεί την Κίνα ή τι Ηνωμένε Πολιτείε. Παρ' όλα αυτά, η πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους περιορίζει, καθιστά την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασθενέστερη και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η Κομισιόν οφείλει να αναγνωρίσει ότι η πολιτική ανταγωνισμού δεν είναι απλά και μόνο ένα νομικό ε, χρηματοοικονομικό εργαλείο. Αν αποτύχει, είναι πολύ δυσάρεστο και αποκόπτεται ε, από την πραγματικότητα. Διερωτώ με κατά πόσο η Γενική Διεύθυνση Αρμόδια κοιτάει και πέρα από την Ευρώπη. Αν αυτό δεν ισχύει, τότε οι απόψει τη ίσω έχουν είναι πολύ αυτιστικές. Ε, πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στο trickle down η θεσπόσα θέση εξαρτάται και από το πώς ακριβώς ορίζεται. Μεταθέτοντας τον ορισμό, ανοίγουμε τις πόρτες ε, στο, στις καταχρήσεις. Η Microsoft ποτέ θα μπορέσει να πετύχει στην Ευρώπη, διότι η Ευρωπαϊκή Πολιτική Ανταγωνισμού ε, θα την είχε κατακρεουργήσει. Ε, γι' αυτό λοιπόν δεν πρόκειται για ευρωπαϊκή εταιρεία, πρόκειται για αμερικανική. Όμως αυτό είναι υποφελές στους καταναλωτές όλου του κόσμου. Αυτό το trickle down effect και ο καταναλωτής, η έννοια της δεσπόσας θέσης, όλα αυτά πρέπει να εκτεστούν σε βάθος αντί να τα ανάγουμε πάνω σε βάθρο. Κατόπιν όσον αφορά τα πρόστιμα κύριε Πρόεδρε, χρησιμοποιήθηκαν ως φόβητρο προς όλες τις κατευθύνσεις και για αθώους που δουλεύουν σε εταιρείε και χάνουν τη δουλειά τους. Τα πρόστιμα κύριε Πρόεδρε δεν υπάρχουν ε, για να ενισχύουν το κύρος ε, της Επιτροπής ή των Επιτρόπων ούτε υπάρχουν ε, για να καλύπτουν τις τρύπες του προϋπολογισμού πρέπει τα πρόστιμα να επιβάλλονται οποτεδήποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο στους παραβάτες. Γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα η Κομισιόν πρέπει να παραμείνει πιστή στην αποστολή της. Με ένα λογοπαίγνιο το λέει ο μιλητής. Επίσης πρέπει να δούμε τον αγροβιομηχανικό τομέα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στη διάθεσή της ε, κοινή γεωργική πολιτική. Δεν την επικρίνω σε επίπεδο αρχής, όμως γνωρίζω ότι οι μεγάλες αγροβιομηχανικές εταιρείε είναι οι βασικοί αποδέκτες των ενισχύσεων και όχι οι γεωργοί όπως πιστεύουν πολλοί. Βέβαια, οι τιμέ των τροφίμων στην Ευρώπη είναι πολύ ψηλέ. Οι Ευρωπαίοι πολίτε χρηματοδοτούν την ΚΑΠ και τα ωφέλη πηγαίνουν στον αγροβιομηχανικό τομέα. Όμω, ο Ευρωπαίο καταναλωτή πληρώνει υψηλέ τιμέ ε, τροφίμων στην τελική αγορά. Αυτό είναι ανισότητα και πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια σε αυτόν τον τομέα, έχοντας κατά νου ε, τις ε, τελικές ε, τιμές καταναλωτή και καλό την αρμόδια, το αρμόδια Γενική Διεύθυνση Επιτροπής να λάβει τα μέτρα, για τα μέτρα που πρέπει για να υπηρετεί τον Ευρωπαίο καταναλωτή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Θέτει αρκετά ενδιαφέροντα σημεία έχοντας διαβάσει και τα κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την, το σχέδιο έκθεσης του κυρίου Έπιν. Σε τρία σημεία θα σταθώ. Το πρώτο αφορά τον ανταγωνισμό και τις μικρομεσαίες. Είναι σαφές ότι απαιτείται να, να συντάξουμε εκ νέου τους κανόνες ανταγωνισμού που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η δημιουργία θέσεων απασχόλησης ε, ουσιαστικά ε, έχει περιοριστεί σε αυτό το κομμάτι της οικονομικής δραστηριότητας. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά προβλήματα σε σχέση με τις διασυνοριακές ε, κυρίως δραστηριότητες των μικρομεσαίων. Για το θέμα των προστήμων είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα θα πρέπει να συζητηθεί. Τα υψηλά πρόστιμα είναι αποτελεσματικός άραγε τρόπος για να επιβληθεί ο σεβασμός των κανόνων. Μήπως κάποια από τα πρόστιμα αυτά είναι δυσανάλογα ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της κρίσης. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να θέσουμε. Για την αγορά της ενέργειας σε σχέση με τον ανταγωνισμό έχουμε στην Ευρώπη κάποιες δυσκολίες. Δεν εννοώ εδώ τα προβλήματα στη διασύνδεση που έχουμε σε πολλές ε, περιοχές της Ευρώπης αλλά έχουμε διαφορετικά προβλήματα σε σχέση με τους προμήθευτές. Σε ορισμένες χώρες έχουμε διαφορετικά κριτήρια, έχουμε σε, ανάλογα με τη χώρα ε, για το ποιος είναι ε, ένας ε, θα έλεγα πελάτης σε εισαγωγικά εισαγωγέας ο οποίος υπόκειται σε συγκεκριμένους κανόνες ή ένας άλλος ο οποίος υπόκειται σε διαφορετικούς κανόνες αν έχετε τον Τάδε ο οποίος ε, που πολύ ενέργεια σαν παράδειγμα στον Δίνα η ε, συναλλαγή αυτή γίνεται μερικές φορές ε, με μία μη διαφανή λογική και δημιουργεί στρεβλώσεις γενικότερα στην αγορά ενέργειας. Θα πρέπει λοιπόν να υπογραμμίσουμε εδώ ότι οι κανόνες θα πρέπει να γίνουν πιο κατανοητοί, να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει και τι πρέπει μάλλον να συμβεί περισσότερο σε ευρωπαϊκή βάση ξεπερνώντας τις εθνικές διαφορές. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο, έχω την αίσθηση ότι οι προτάσεις του εισηγητή είναι γενικά θετικές. Ευχαριστώ κύριε Κάρινς. Πρεσέδο. Ευχαριστώ πρόεδρε. τα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς και για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας στα πλαίσια της πολιτικής ανταγωνισμού η έκθεση της Επιτροπής έχει συμπεριλάβει δεν έχει συμπεριλάβει κάτι το οποίο θέτουμε εμείς. Δηλαδή υπηρεσίε γενικού ενδιαφέροντο. Νομίζω ότι θα πρέπει το θέμα αυτό να το συζητήσουμε περαιτέρω. Και ίσω αναφορά στου καταναλωτέ γίνεται με πολύ λακωνικό τρόπο. Ούτω ή άλλω υπάρχει ένα ειδικό ε, κεφάλαιο θα πρέπει να υπάρχει ειδικό κεφάλαιο για την χρηματοπιστωτική κρίση, δεδομένου ότι η πολιτική ανταγωνισμού, όπω ξέρουμε, συνεισέφερε πάρα πολύ στην ε, αποκατάσταση τη ε, σταθερότητα δίδοντας ίδιες ευκαιρίες, τι τι ίδιες δυνατότητες όρου και συνεχίζει να παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για την ομαλοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Υπάρχει ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό που συνέβη από πέρσι. Και θα αναφέρω τις συλλογικές Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να το ξεχάσουμε. Σε πολλές, φορ... πολλές φορές ξέρουμε ότι έγιναν δηλώσεις από κάποιες πηγές της Επιτροπής, όχι στα πλαίσια του ανταγωνισμού, αλλά σε άλλα θέματα που είναι κάπως συγκεχημένες. Σε σχέση λοιπόν με την αποδοτικότητα της ε, ε πολιτικής ανταγωνισμού θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα πρόστιμα και οι κυρώσεις που επιβάλλονται. Πάντα βεβαίως θα πρέπει να έχουν αποτροπτικό χαρακτήρα. Διαφορετικά η πολιτική ανταγωνισμού θα δημιουργεί κίνητρα ε, κατά του υγιούς ανταγωνισμού. Υπάρχουν ε, προτάσει εδώ που συμπεριλαμβάνονται και είναι σωστέ. Θα θέλαμε επίση να υπογραμμίσω σημαντική είναι η πολιτική αυτή στα πλαίσια των ΜΜΕ, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κατά την άποψή μα τα θέματα που είναι επίση πολύ ενδιαφέρονται, αυτά που αφορούν την διατροφική ε, αλυσίδα. Νομίζω ότι όταν ολοκληρώνουν τι εργασίε του τα μέλη τη ομάδα υψηλού επίπεδου θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα πορίσματα τα οποία θα συνάγουμε και θα προσπαθήσουμε με εμεί με επικοδοτικό τρέμα πνεύμα να καταθέσουμε και τροπολογίε για να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια νέα όθηση στην πολιτική ανταγωνισμού. Δηλαδή, <coughs> Ευχαριστούμε κύριε Σάντσες. Η κυρία Ήμπελ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ξεκινώντας θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον Έπινγκ. Νομίζω ότι μπορούμε όλοι να δούμε ότι εγώ που ήμουν περσινή συγγήτρια βρίσκω πάρα πολλά κοινά σε αυτά τα οποία είπε. Μια γενική υποκαταρτική παρατήρηση. Έχω την εντύπωση ότι πέρυσι έγινε μια αντίστοιχη συζήτηση και είναι προφανές ότι και τον προπροηγούμενο χρόνο πάλι η συζήτηση ήταν παρόμοια και φοβάμαι ότι για μια ακόμη φορά θα συζητήσουμε τα ίδια πράγματα. Ένα από τα βασικά θέματα τα οποία έθεσα πέρυσι είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη αυτά τα οποία ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είχαμε θέσει συγκεκριμένες ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είχαμε ζητήσει εκθέσεις, είχαμε ζητήσει αναλύσεις και δεν πήραμε απολύτως τίποτα, ούτε καν μια συνοπτική απάντηση. Λοιπόν, δεν θέλουμε ευγενικά λόγια από πλευρά του Επιτρόπου. Θέλουμε ε, όταν ζητάμε απαντήσεις να μας δώσει απαντήσεις. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει να δώσει απαντήσεις, να το πει να πάνε και αυτοί και εμείς στα σπίτια μας να πιούμε ένα τσαγάκι και να ηρεμήσουμε όλοι. Λοιπόν, πρέπει να συνειδητοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει και σε πάρα πολλούς ε, τομείς της πολιτικής μας τα πράγματα είναι διαφορετικά από ό,τι πριν μερικά χρόνια. Γιατί αυτό. Γιατί θέλουμε οι αποφάσεις της, Ευρωπαϊκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λαμβάνονται με μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμοποίηση. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα φανεί σοφή θα έλεγα λαμβάνοντας υπόψη επιτέλους τις απόψεις του άμεσα εκλεγμένου Δημοκρατικού Σώματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές βοήθειες. Επαναλαμβάνω αυτά τα οποία είπα πέρυσι. Έχουν δοθεί τεράστια ποσά σε πάρα πολλούς τομείς τα τελευταία χρόνια. Για πάρα πολλά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε καταφέρει να μειώσει τα ποσά αυτά τα κρατικά. Παρ' όλα αυτά τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει η κατάσταση. Εμείς θα θέλαμε τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων να δαπανώνται με σωστό τρόπο. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση παίρνουμε εκθέσεις ε, για το ποιες αποφάσεις έχουν ληφθεί και σε ποιες περιπτώσεις, αλλά δεν παίρνουμε εκθέσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις επιπτώσεις αυτών των ε, βοηθειών, των επιδοτήσεων. Σαν παράδειγμα, η πράσινη ανάκαμψη, οι κρατικές βοήθειες έχουν βοηθήσει καθόλου. Έχουμε προχωρήσει στην ε, λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη, ανάκαμψη της οικονομίας ή χάνουμε και εκεί λεφτά. Λοιπόν, απαντήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δίνει απαντήσεις. Όταν θέτουμε ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ανταποδίδει ωραία χαμόγελα και απόλυτη σιωπή. Έχω ζητήσει σαν παράδειγμα μία έρευνα σε συγκεκριμένους τομείς όπως ε, η έρευνα. Γιατί δεν παίρνω απάντηση ποτέ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν δεν θέλει να δώσει απάντηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ας το πει επιτέλους. Τώρα για τα μέτρα αντιτράστ. Νομίζω ότι και πέρυσι είχαμε ζητήσει να μας δοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια ανακοίνωση επίσημη και μια πρόταση γενικότερα παρουσίασης των προβλημάτων που έχει ας το σύστημα επαβολής, επιβολής προστήμων. Έτσι ώστε να δούμε ακριβώς τι ρόλο μπορεί να παίξει. Λοιπόν, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε κάνει αυτή την ανακοίνωση και είχε κάνει προτάσεις θα είχαμε μια σωστή βάση για συζήτηση κάτι το οποίο δεν έχουμε δυστυχώς. Λοιπόν μπορούμε να συζητάμε εμείς, να παίρνουμε αποφάσεις, να ψηφίζουμε, να καταθέτουμε τροπολογίες, να γνωστοποιούμε την άποψή μας. Το θέμα είναι αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αρχίσει να μας λαμβάνει υπόψη. Αν δεν το κάνει αυτό τότε γιατί συζητάμε. Ευχαριστώ. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό το οποίο είπε η Σοφή. Όπως έλεγε ένας Ισπανός φιλόσοφος, η ανώφελη προσπάθεια, η άχρηστη προσπάθεια οδηγεί στη μελαγχολία. Συμφωνώ λοιπόν με αυτά που είπε η Σοφή. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο για να αντιδράσω στις παρατηρήσεις που έγιναν. Συμφωνώ ότι πρέπει να ασχοληθούμε με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πολύ σημαντικό. Και επίσης να πω ότι η οδηγία περί υπηρεσιών και αυτή είναι πολύ σημαντική, διότι έχουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που υποφελούνται από διασυνοριακές δραστηριότητες. Άρα η σωστή εφαρμογή της οδηγίας περί υπηρεσιών είναι πολύ σημαντική και αυτό εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς. Τέλος, όσον αφορά τις αγορές ενέργειας και εκεί συμφωνούμε, πράγματι οι πολίτες καταβάλουν ε, υψηλά ποσά για την ενέργεια. Δεν υπάρχει κατ' ουσίαν ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Συμφωνώ, και με αυτό. Και με αυτό που πρότεινε ο κύριος Σάντσες ε, σχετικά με την εξέλιξη τιμών ε, στον τομέα των τροφίμων. Είναι σημαντικό να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για να προστατεύσουμε τον καταναλωτή διότι όπως σας είπα οι καταναλωτές ε, πληρώνουν διπλάσεις τιμές. Πληρώνουν για την ΚΑΠ και πληρώνουν και για τις υψηλές τιμές τροφίμων. Άρα δηλαδή κάτι δεν πάει καλά. Κύριε Ιντφέλτ, ε, πραγματικά ζηλεύω ε, τον ζήλο σας και την στράτευσή σας για το τον αγώνα σα με την ε, Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Το έκανα και εγώ παλιά και αυτό που μου έμεινε το εξή ότι ο ανταγωνισμός είναι η ιερή αγελάδα. Οι επίτροποι κατά κανόνα δεν παρεμβαίνουν σε αυτά που λέει ή κάνει ο Επίτροπος, Επίτροπος Ανταγωνισμού. Ο Επίτροπος Ανταγωνισμού συμφωνεί ε, με τον πρόεδρο της Επιτροπής και το θέμα έκλεισε. Κανείς πια δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ε, η μόνη διαμαρτυρία μπορεί να γίνει από το κράτος μέλος και αυτό μόνο για τα πρακτικά. Έτσι λοιπόν ε, θεωρώ ότι η τρέχουσα πολιτική ανταγωνισμού δεν συμβαδίζει με τα τεκτενόμενα ανά τον κόσμο. Είναι απομονωμένη, αποκομμένη. Είναι μια έννοια που λειτουργεί αυτόνομα. Ξεχνάει όμως το τι συμβαίνει γύρω της. Κυρίως ε, αγνοεί τις ε, τάσεις ανά τον κόσμο. Φοβάμαι λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή η πολιτική ανταγωνισμού υπονομεύει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που δεν είναι σε θέση να ανταγωνιστούν σε διεθνές επίπεδο. Πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα ευρύ πνεύμα, μια ευρία συζήτηση εδώ στο Κοινοβούλιο καλούμεθα να αναγκάσουμε την ε, ε, Κομισιόν ε, να φύγει από αυτό το γυάλινο πύργο μέσα στον οποίο είχε βολευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η κυρία Ινεφέλ και εγώ θα συνεχίσουμε με τη συζήτηση και σας ευχαριστώ πολύ για όλες. Η συζήτηση θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα. Ζήτησε το λόγο η Επιτροπή, έχουμε χρόνο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you very much. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον εισηγητή για αυτό το σχέδιο ψηφίσματος ε, που θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα περιεκτικό και το οποίο θίγει πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Ε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να απαντήσω στο γενικότερο αίτημα που υποβλήθηκε στην Κομισιόν ότι η Κομισιόν δεν ε, ανταποκρίνεται στις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει να σας πω, χαιρετίζουμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι η ψηφοφορία για το ψήφισμα προτάχθηκε κάτι που θα μας επιτρέψει εμείς να λάβουμε υπόψη μας το ψήφισμα όταν θα δημοσιεύσουμε την ετήσια έκθεση ε, περί ανταγωνισμού. Αυτό λοιπόν είναι μια θετική εξέλιξη και θα μας ε, επιτρέψει να δώσουμε και εμείς ε, μια ικανοποιητική απάντηση στο έτοιμά σας. Όσον αφορά στο συγκεκριμένο θέμα για το ψήφισμα της ε, περασμένης χρονιάς, θέλω να πω ότι εμείς στείλαμε μια λεπτομερή απάντηση στο Κοινοβούλιο, στον πρόεδρο της ε, Επιτροπής της Οικονομικής και βεβαίως ε, και στα μέλη μετά από αίτημα της Πρόεδρου. Άρα δηλαδή θα ήθελα παρακαλώ και αυτό ή δυνατόν να το αναγνωρίσετε. Όσον αφορά τώρα γενικότερα την ουσία της έκθεσης, εμείς ε, χαιρετίζουμε την ευρύτερη υποστήριξη προς την πολιτική ανταγωνισμού. Ε, λαμβάνουμε υπόψη μας το γεγονός ότι η έκθεση σε μεγάλο βαθμό ε, δίδει σημασία στον έλεγχο των ισχύσεων και στην πολιτική ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια κρίσεων. Πολύ σωστό αυτό. Και όπως και πολλοί ανέφεραν εδώ, η πολιτική ανταγωνισμού είναι ένα αναπόφευκτο εργαλείο για να διασφαλίζουμε ίσους όρους ανταγωνισμού ε, με τους ε, εταίρους μας ανά τον κόσμο. Όσον αφορά το προσωρινό πλαίσιο και τις ε, ανησυχίες που εκφράστηκαν ότι ίσως τελικά το προσωρινό να είναι και μόνιμο, να μην είναι και τόσο προσωρινό, εγώ θέλω να πω ότι αυτό το προσωρινό πλαίσιο πράγματι εκπνέει ε, στο τέλος του έτους. Η Κομισιόν θα συγκεντρώσει, θα αναλύσει όλες τις πληροφορίες για την ε, χρησιμότητα του προσωρινού αυτού πλαισίου. Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε όλες τις ε, απαντήσεις που λάβαμε μετά από διαβουλεύσεις. Θα αναλύσουμε ενδελεχώς αυτές τις απαντήσεις την επόμενη εβδομάδα στις 5 Οκτωβρίου. Ο Αντιπρόεδρος κ. Αλμούνια θα έρθει εδώ και θα απαντήσει ε, σε όλες σας τις ε, ερωτήσεις επ' αυτού του θέματος. Τώρα, ε, θα ήθελα να αναφερθώ και στις απόψεις που εκφράστηκαν για την πολιτική μας κατά των τραστ και των συγχωνεύσεων, κυρίως για τα πρόστιμα. Να υπογραμμίσω ότι τα πρόστιμα επιβάλλονται για να προστατευθεί το δημόσιο συμφέρον. Και έχουν ένα στόχο που είναι ανεξάρτητος ε, από ε, τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το οποίο κάπως υπονοεί το ψήφισμα. Δηλαδή τα πρόστιμα ε, που δεν είδαν επιβάλλονται για να τροφοδοτήσουν τον κοινοτικό προπολογισμό. Σωστό, κατευθύνονται προς τα εκεί, αλλά μετά επιστρέφονται πίσω στα κράτη-μέλη ανάλογα με τη συνεισφορά τους. Άρα δηλαδή με αυτή την έννοια τα πρόστιμα είναι ουδέτερα στις επιπτώσεις τους. Εμείς βεβαίως και εξετάσαμε τις διάφορες προτάσεις για τη σημασία των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης λάβαμε υπόψη μας τις παρατηρήσεις που έγιναν για τα τρόφιμα. Εγώ θα ήθελα απλά να υπογραμμίσω κάτι που αφορά στην ενέργεια, όπου ο εισηγητής ε, εκφράζει τη δυσαρέσκειά του και άλλοι για την κατάσταση που επικρατεί στα κράτη-μέλη. Να πω λοιπόν ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει να είναι ιδιαίτερα αυστηρή στο να εφαρμόζει τους κανόνες ανταγωνισμού στην ενέργεια, κυρίως σε περιπτώσεις κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης στον τομέα της ενέργειας, όπως συμβαίνει και με το ηλεκτρικό ρεύμα και το αέριο. Οι εξελίξεις έχουν οδηγήσει στον να μεγαλύτερη ασφάλεια ανεφοδιασμού, ε, προσθέσει του περιβάλλοντος, μεγαλύτερες καινοτομίες ε, και ε, παροχή ενέργειας σε ανταγωνιστικές τιμές για τα νοικοκυριά και για τις εταιρείες. Και θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μου έστειλε απάντηση σε μένα, ε, την εισηγήτρια και τον Πρόεδρο. Εγώ δεν πήρα καμία προσωπική απάντηση. Βρήκα μία απάντηση εδώ και αρκετούς μήνες που δεν ήταν απάντηση. Ήταν ουσιαστικά η περίληψη των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την ανάλυση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών σας. Ίσως για σας να φαίνεται μια επιστημονική, εμπάση περιπτώσει, επανάσταση, αλλά πράγματι όταν παίρνετε κάποιες αποφάσεις δεν είναι αυτός σκοπός. Πρέπει να προσμετρήσετε τις επιπτώσεις. Αν δεν προσμετρήσουμε τις επιπτώσεις και τις συνέπειες των δισεκατομμυρίων κρατικών επιδοτήσεων, τι θα καταλάβουμε αν ήταν χρήσιμες ή όχι ή αν θα πρέπει να παραταθεί σαν παράδειγμα το προσωρινό πακέτο, το οποίο δεν φαίνεται να είναι και τόσο προσωρινό. Πού θα βασίσετε την απόφαση αυτή. Έχετε κάνει κάποια μελέτη για τις επιπτώσεις των επιδοτήσεων. Σε ποιο βαθμό σαν παράδειγμα έχει πετύχει τους στόχους που είχατε θέσει. Και είχαμε κάνει αρκετές προτάσεις σε ποιου ιδιαίτερα τομείς θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει κάποιες μελέτες και δεν πήραμε απάντηση. Δεύτερη ερώτηση που μπορείτε να μου απαντήσετε ναι ή όχι. Θα υπάρξει ε, θα υπάρξουν οι έρευνες αυτές οι τομεακές τις οποίες έχουμε παραγγείλει, έχουμε ζητήσει. Commission, please. Επιτροπή Σχετικά με τις επιπτώσεις των πολιτικών μας αποφάσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογεί, εν πάση περιπτώσει, πριν ξεκινήσει ε, μια νέα νομοθετική δραστηριότητα και πάρα πολύ πιθανώς, αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο ο πρόεδρος Μπορόσο έχει ζητήσει από πέρυσι, μια αξιολόγηση των υστέρων των πολιτικών αυτών. Είναι αλήθεια ότι στο παρελθόν η πολιτική ανταγωνισμού που ήταν μια θα έλεγα πολιτική επιβολή συγκεκριμένων μεθόδων και αποφάσεων δεν οδηγούσε σε αξιολογήσεις εκ των υστέρων. Παρατηρείται όμως ότι οι περισσότερες από τις νέες κατευθυντήριες γραμμές, όπως οι οριζόντιες κατευθυντήριες γραμμές, περιλαμβάνουν μελέτες επιπτώσεων και αυτό θα συνεχιστεί στο μέλλον και στον τομέα των κρατικών βοηθειών. Πριν λοιπόν εμείς ε, προχωρήσουμε στις μελέτες επιπτώσεων θα ε, προχωρήσουμε και ε, στις αξιολογήσεις που προαπαιτούνται δεν έχουμε δυσκολίες όταν προσπαθούμε φυσικά μερικές φορές να αξιολογήσουμε και να προσμετρήσουμε τις επιπτώσεις των πολιτικών ανταγωνισμού και στον τομέα των κρατικών βοηθειών και σε άλλους τομείς. Αλλά προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό, όχι μόνο επειδή μας ζητείτε, αλλά γιατί έτσι είμαστε πραγματικά υπόλογοι απέναντι στα πολιτικά, σχετικά με τις τομεακές έρευνες που ζητήσατε. Αυτή είναι μια απόφαση την οποία ο Αντιπρόεδρος ε, Αλμούνια θα πρέπει κάποια στιγμή να πάρει. Λοιπόν, ο εισηγητής θέλει να κάνει κάποια τελική παρατήρηση. Έπινγκ. Νομίζω ότι αυτά δείχνουν ότι πράγματι ε, έχουμε ανάγκη την ακρόαση της εβδομάδας της επόμενης. Ελπίζω να είναι η κυρία Ιντβέλτ ελπίζω να ψήσουμε τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Θυμάμαι κάτι που είχε πει ο Φίλιπ Λόου, ότι η τότε επίτροπος η κυρία Κρούζ έκανε ό,τι της έγραφε η γενική της διεύθυνση. Ελπίζω να αλλάξει η κατάσταση με τον κύριο Αλμούνια τώρα. Γιατί αν ο επίτροπος λέγει μόνο αυτά που του γράφουν οι υπάλληλοι του, τότε αυτό σημαίνει ότι η γραφειοκρατία είναι το αφεντικό σε αυτή την υπόθεση. Και τότε η πολιτική ανταγωνισμού θα ξεφύγει από τον πραγματικό κόσμο. Γι' αυτό ακριβώς θα κάνουμε την ακρόαση την επόμενη εβδομάδα και θα τα θέσουμε με πολύ ομό τρόπο αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε και η συζήτηση για το θέμα αυτό. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, θα σας εξηγήσω. Προθεσμία Προθεσμία τροπολογιών, 7 Οκτωβρίου, μέχρι τις 5 το απόγευμα. Συζήτηση στις 26 Οκτωβρίου ψηφοφορία στην Επιτροπή μας 30 Νοεμβρίου και ολομέλεια στην 1η Δεκεμβρίου. Συμφωνεί ο εισηγητής, εάν ναι, έληξε η συζήτηση, στα διάφορα θέλει κανείς να προσθέσει κάτι, εάν όχι, λύεται η συνεδρίαση. Αν θέλει ο Θεός, θα ξανασυντοντηθούμε στις 3 ώρα το απόγευμα τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου.